Care collega, cari colleghi, dichiaro aperta Αγαπητοί συνάδελφοι, άρχεται η συνεδρίαση της διάσκεψης των Προεδρών που είναι ανοιχτή σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Καταρχάς, θέλω να ζητήσω συγγνώμη εξ ονόματος του Πρόεδρου Σούλτς για την απουσία του που οφείλεται σε μια ε, δυνατή γρήπη. Νομίζω ότι εξ ονόματος όλων θα ήθελα να εκφράσω τις ευχές ε, για ταχύ ανάρρωση προς τον Πρόεδρο. Δεύτερον, να καλωσορίσω τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Βαν Ρομπάη και τον Πρόεδρο της Επιτροπή κ. Μπαρόζο και όλους σας. Κύριε Πρόεδρε Βαν Ρομπάη, πριν σας δώσω το λόγο, να συνεχίσω. Κύριε Ντί, Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνουμε την ιδιαίτερη κατάσταση της Ένωσης, αλλά βάσει του άρθρου 15.6 δέλτα της συνθήκη θέλω να ρωτήσω τι αντιτίθεται στο να λογοδοτήσει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο σώμα ολόκληρο και όχι στη διευρυμένη διάσκεψη των Πρόεδρων. θυμάστε κύριε Πρόεδρε ότι το είχα σχολιάσει αυτό το θέμα ήδη. Είναι διαφορετική η Ολομέλεια από την διάσκεψη των Πρόεδρων και ως προς τη δημοσιότητα το δικαίωμα των ε, βουλευτών να λάβουν το λόγο και αλλάζει την κατάσταση για ιστορικούς, για τους πολίτες, Ρωτώ λοιπόν γιατί ο πρόεδρος του Συμβουλίου δεν θέλει να έρθει ενώπιον του Κοινοβουλίου και, και επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν έχει να κάνει, ότι δεν έχει να, η παρέμβασή μου να κάνει τίποτα με την ε, ιστορία του κτηρίου εδώ στο, στις Βρυξέλλες. Είναι ένα θεσμικό ζήτημα που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πολύ ισχυρούς λόγους για να μας πει, να σας εξηγήσει ο πρόεδρος γιατί δεν θέλει να μιλήσει ενώπιον ε, της ολομέλειας. Ευχαριστώ κύριε ότι Έχετε δίκιο θεωρητικά. Αλλά πρέπει να είστε και ρεαλιστέ. Αν θέλαμε να περιμένουμε την επόμενη ολομέλεια για να έχουμε μια ενημέρωση για το Συμβούλιο, θα περιμέναμε το Στρασβούργο. Πολύ αργά. Εμείς αντίθετα χρειαζόμαστε να ακούσουμε και να αντιδράσουμε σε αυτά που θα πει ο πρόεδρος κ. Βαν Ρομπάη και χρειάζεται τούτο να γίνει Γνωρίζετε ο... και εσείς και εμείς ότι δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουμε την έφυση της Ολομέλειας της Βρυξέλλες και για το λόγο αυτό η διάσκεψη των πρόεδρων ανοιχτή σε όλα τα μέλη είναι ανοιχτή με πρακτικά και μπορεί ο καθένας να τα παρακολουθήσει. Πριν δώσω το λόγο στον πρόεδρο Βαν επιτρέψτε μου να εκφράσω την απογοήτευση, ένα αίσθημα απογοήτευσης που ε, κυριαρχεί Εβραίος στο Κοινοβούλιο και που εκφράστηκε από δημόσιες δηλώσεις των πρόεδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων και από τον ίδιο τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Απογοήτευση προκύπτει από το γεγονός ότι η συμφωνία που επιτέθηκε στο Συμβούλιο δεν μας φαίνεται στο ύψος των προκλήσεων που μας αναμένουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε και συνεχίζει νομίζω να ζητά ένα σύγχρονο και φιλόδοξο προπολογισμό ικανό να υποστηρίξει την ανάκαμψη της Ευρώπης και να συμβάλλει το να θέσουμε πίσω πλέον την οικονομική, κοινωνική και χρηματοοικονομική κρίση. Μακράν είμαστε τις προσδοκίες αυτής και είναι κρίμα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι δύσκολο να, αδύνατο να αντιμετωπίσουμε μια δυσκολία οικονομική εν ώψη αυτής της μείωσης του προπολογισμού. Αποτελεί τούτο ένα βήμα πίσω που δεν θα είχε καμία λογική και δεν μπορεί να είναι κατανοητό το ούτε από εμά ούτε από του Ευρωπαίου πολίτες. Σε μια στιγμή που ξεκινούμε να βλέπουμε τα πρώτα δειλά ε, μηνύματα της ανάπτυξης θα ήταν λογικό να επενδύσουμε στην Ευρώπη και να ε, προχωρήσουμε σε βασικές ε, αλλαγές της ευρωπαϊκής πολιτικής τις πολιτικές της Ευρώπης για την επόμενη δεκαετία. Έρευνα, ανάπτυξη, εξωτερική πολιτική, ε, πολιτική ανάπτυξη. Μια τέτοια συμφωνία κύριε Πρόεδρε δεν είναι προς το συμφέρον του Ευρωπαίου πολίτη. Οι περικοπές που προτείνεται θα έχουν ε, σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και για το λόγο του αυτό το κοινοβούλιο θα μπορέσει να δεχθεί τη συμφωνία ως έχει. Το λόγο έχει ο αξιότιμος πρόεδρος κ. Βαν Ρομπάη. Κύριε Πρόεδρε, εξότιμοι κυρίε και κύριοι, στις 7 και 8 Φεβρουαρίου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών κατέληξαν σε συμφωνία στο δικό τους επίπεδο για το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης στις προσεχούς 7 ετίας. έχουν ελαφρώς μειωθεί σε σχέση με, το προηγούμενο, με την προηγούμενη εφταετία τα ε, όρια, αλλά μέσα στο πλαίσιο αυτό έχει αλλάξει και η σειρά των προτεραιοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται λοιπόν στις ε, ε επενδύσεις στην ανάπτυξη της εργασίας. Έτσι ικανοποιούνται δύο βασικές, η βασική επιλογή του με δεδομένες τις περικοπές τους προϋπολογισμούς στην Ευρώπη και τη λιτότητα να επενδύουμε στο μέλλον. Από την, ε, τις αναφορές του τύπου κάθε επικεφαλής, κάθε αρχηγός κρατός και κυβερνήσεως προσπάθησε να κερδίσει όσο περισσότερα πλεονεκτήματα δυνατά για τους πολίτες του. Θεμητό, θεμητό στόχος, δεδομένου βέβαια ότι ορισμένοι επικεντρώνονται περισσότερο στον φορολογούμενο και άλλοι στον δικαιούχο. Για μένα σημαντικό ήταν να καταλήξουμε από κοινού σε μια συμφωνία, σε μια καλή για την Ευρώπη συνολικά συμφωνία. Χρειάστηκε να αναζητήσουμε συμφωνία επί τριών παραμέτρων. Το μέγεθος, τον όγκο δηλαδή, τις προτεραιότητες των δαπανών και τις πηγές των ε, εσόδων. Με επιδίωξη έναν εξυγχρονισμένο και εστιασμένο προπολογισμό, κυρίως για τις πιο επίγουσες ανάγκες. Ως προς τον όγκο λοιπόν, ως προς τα μεγέθη, με δεδομένες τις τωρινές ε, δυνατότητες, ο προπολογισμό ήταν ε, βέβαια μετριοπαθής, σφίγγουν τα ζωνάρια σε όλη την Ευρώπη και η Ένωση δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Ορισμένοι θεώρησαν ότι κατά 3% ε, μείωση του, το 3% για τις δεσμεύσεις υποχρεώσεων ήταν ε, πολύ αυστηρή. Ωστόσο, σε ολόκληρη την Ευρώπη προσπαθούμε να κάνουμε στο δυνατόν περισσότερα με λιγότερα κονδύλια, ώστε να μπορέσει το κάθε ευρώ να αποδίδει το μέγιστο. Περισσότερη Ευρώπη δεν συνεπάγεται απαραίτητα και περισσότερα κονδύλια. Αλλά θα ήθελα επίση να υπογραμμίσω ότι στι δεσμεύσει υποχρεώσεων η μείωση αυτή μπορεί να μην έχει και συνέπεια για τι πραγματικέ πληρωμέ στου ετήσιου προπολογισμού που θα εγκρίνετε εσεί. Στην τελευταία, τελευταία επτά αιτία οι πληρωμέ που ενέκρινε το Κοινοβούλιο ήταν πολύ χαμηλότερες από το το όριο του ε, πολιτού δημοσιονομικού ε, πλαισίου και έφτασαν στα 874 δισεκατομμύρια, πολύ λιγότερα δηλαδή από τα 908 που προβλέπονται για, το προσεχές, για την προσεχή επταετία. Τα Ανώτατα όρια λοιπόν του δημοσιονομικού πλαισίου δεν θα μπορούσαν ούτε προ τα πάνω ούτε προ τα κάτω να μειωθούν παρά μόνο για ολίγε ποσοστιαίε μονάδε και δεδομένε και τη ανάγκη τη ομοφωνία. Πάντω κάποια ε, οικονομικά σχόλια επικεντρώνονται μόνο στην πτυχή αυτή, τη μείωση δηλαδή. Ε, θα ανατρέξω στο Νοέμβριο όπου εγώ προσωπικώ είχα υποβάλει μια συνολική πρόταση για 917 δισεκατομμύρια, για για 970 ε, και τα 960 εκατομμύρια ήταν σχετικά κοντά, αν και κάποια, ε, κάποια θέλανε να μειώσουν κατά 30 δις ή περισσότερο ακόμη τη δική μας αρχική πρόταση. Εάν λοιπόν ρίξουμε μια ματιά τώρα στο περιεχόμενο, το δεύτερο σημείο των δαπανών. Εδώ βλέπουμε σημαντικές αλλαγές για τις οποίες αξίζει να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας. Η σημασία αυτών των αλλαγών στάθμισης είναι πολύ μεγαλύτερη από την ε, σχετικά μικρή περικοπή στο, στη συνολική περικοδότηση και αξίζουν περισσότερης προσοχής αυτές οι αλλαγές. Πρώτον, στο κεφάλαιο 1α, στην κατηγορία 1α, έρευνα, καινοτομία, διασυνοριακή ενέργεια, μεταφορές, ψηφιακά δίκτυα. Γαλιλαίος Εράσμους. Αυτή η κατηγορία βλέπει αύξηση 37,3% σε σχέση με το προηγούμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, 37,3% αύξηση στην κατηγορία 1α. Επιπλέον, η αύξηση αυτή ε, έχει παρουσιάσει και μια χαρακτηριστική σταθερότητα με συνολικό 40% αύξηση στο τέλος της ε, περίοδου. Δεδομένης τώρα της κατάστασης που έχουμε αυτή τη στιγμή, σημειώνεται σημαντική βελτίωση Βεβαίω μπορεί κανεί να εκφράζει τη λύπη του για το ότι δεν έγιναν δεκτέ όλε οι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι επενδύσει, αλλά θα ήταν παρερμηνία της κατάστασης το να παρουσιάζονται ως περικοπές αυτές οι διαφορές, ενώ ουσιαστικά έχουμε περισσότερα κονδύλια για τις επενδύσεις προς την ανάπτυξη από όσα μας έδινε το, μέχρι τώρα που δουπού πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δεύτερον, ε, δαπάνες για τη συνοχή, στι οποίες έχουμε καλύτερη αισθήση και ως εκ τούτου καλύτερα αποτελέσματα, κονδύλια δε ιδιαίτερα αφιερωμένα στις ε, υψηλότερες επιδόσεις θα είναι το χαρακτηριστικό. Με συνεργητική δράση μεταξύ της ε, συνοχής και των, κυβερνητικών, ε, των κρατικών δηλαδή δαπανών. Εν γέννη θα έχουμε πιο απλή αλλά και καλύτερο έλεγχο της διαχείρισης και διαχείριση των κονδυλίων αυτών. Θα ευνοϊκή μεταχείριση στο φόρο προσθέμενης αξίας που θα μπορούν ε, να ε, θα μπορεί να βοηθήσει ως μέτρο τα ε, κράτη της συνοχής. Τα πιο φτωχά κράτη θα έχουν υψηλότερο μερίδιο από την συνοχή, τη χρηματοδότηση της συνοχής, γιατί η συνοχή δεν έχει το βλέμμα στραμμένο προς τα πίσω ως πολιτική, είναι μια επένδυση για το μέλλον. Και επιπλέον υποστηρίζουμε τους πιο αδύναμους, τους πιο φτωχούς, κατά τρόπο σταθερό. Τρίτον, δεδομένη και της αύξησης της ανεργίας των νέων, που επηρεάζει συνολικά έναν στους τέσσερις νέους της Ευρώπης, σε ορισμένε χώρε έναν στου δύο μάλιστα, μια νέα πρωτοβουλία με 6 δισεκατομμύρια ευρώ πρικοδότηση θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση τη τραγική αυτή κατάσταση και αποτελεί, πιστεύω, χαρακτηριστικό παράδειγμα τη κοινωνική διάσταση αυτού του προπολογισμού. Τέταρτον, στην γεωργία. Ε, πρόκειται για ένα πεδίο πολιτική που χρηματοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με επικέντρωση όλο και περισσότερο στην ποιότητα ζωή στην ύπεθρο, πιο πράσινε οικολογικέ δηλαδή δραστηριότητε και αηφόρα παραγωγή τροφίμων. Πολύ μεγάλη σημασία για τους πάντες. Η γεωργία δεν είναι το παρελθόν. Εδώ έχουμε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις στην γεωργική πολιτική που μειώνουν σε ένα βαθμό το σχετικό της ειδικό, το ειδικό της βάρος λες, στον ευρωπαϊκό προπολογισμό με μειωτικές τάσεις. Στον πρώτο λοιπόν πυλώνα της κοινή γεωργικής πολιτικής θα έχουμε περίπου 27% του συνολικού προϋπολογισμού για το πρώτο έτος, πολύ, σημαντικό, ε, πολύ σημαντική μείωση σε σχέση με το 75% που αντιστοιχούσε, όπου αντιστοιχούσε στη δεκαετία του 70 η Γεωργία. Πέμπτον, δαπάνες για την ασφάλεια και την ηθαγένεια. Εδώ βλέπουμε αύξηση 27% γιατί πρόκειται για ένα πεδίο ενισχυμένη και ενισχυόμενη διαρκώ συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Έκτον, εξωτερικές σχέσεις, εξωτερική δράση δεν την παραμελήσαμε και εδώ έχουμε αύξηση 3,3% σε πραγματικούς όρους. Επιπλέον δε δεσμευόμεθα να τηρήσουμε τους, ε, τις δεσμεύσεις μας για τους στόχους της χιλιετηρίδας και στρατευόμεθα σε στόχους ε, παγκόσμιους όπως η ανάπτυξη, όπως η προστασία από τις κλιματικές αλλαγές το Ταμείο Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωση, αντίθετα από ό,τι έχω δει να καταγράφεται στον τύπο, δεν, και υπογραμμίζω, δεν περικόπτεται, του αντίον ενισχύεται. Έβδομον. Ακόμη και στη διοίκηση βλέπουμε μια μικρή ανάπτυξη στο σχετικό, σχετική κατηγορία, γιατί πρέπει να προβλεφθούν οι μεταβολές που θα επιφέρει η διεύρυνση με νέα κρατημέλη. έτσι καταγράφονται ταυτόχρονα σημαντικές, ε, μάλλον σε αυτό θα ενταχθούν και σημαντικές προσπάθειες ε, του προσωπικού για μείωση και σε αριθμούς και, σε, και αντίστοιχα αύξηση χρόνου εργασίας και ε, σε μια παράταση του ορίου σταξιοδότησης με στόχο να έχει πάντα πολύ αποτελεσματική ε, ε, πολύ, αποτελεσματικό προσωπικό στη δημόσιε υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι ήταν σαφή ότι κάποιε αμφιβολίε ε, ορισμένων που είχαν εκφραστεί απαντώνται ικανοποιητικά. Εδώ πρέπει να επισημάνω, περνώντα την επόμενη παρατήρηση, ότι συνήθω μιλάμε για ιδίου πόρου, όπω λέμε, δηλαδή συλλογή από δασμού, από ειδικού φόρου και ε, προσπαθούμε να ενισχύσουμε το ποσοστό των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναζητούνται δε και νέοι ήδη πόροι, παραδείγματι μέσω ενός νέου συστήματος ΦΠΑ και μελλοντικού φόρου των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν επίσης ιδίου πόρου, και έχουμε καταλήξει σε μια συμφωνία ως προς το πολύ δύσκολο ζήτημα της επιστροφής για ορισμένα κράτη. Επιτρέψτε μου επίσης αγαπητοί συνάδελφοι να αναφερθώ σε κάποιες επιμέρους ε, κατηγορίες που απευθύνθηκαν σε αυτήν την ε, συμφωνία καταγράφει αυτή τη συμφωνία, ιδιαίτερα όσον αφορά τι αποκλήσει μεταξύ τη μέσων υποχρεώσεων και πληρωμών. Εδώ Πρέπει να πω ότι βρίσκουμε αντιστοιχεί μετά όσα είχαν συμβεί με το προηγούμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, ωστόσο κάνουμε μια προσπάθεια επιπλέον για να καλύψουμε το χάσμα. Συμφωνούμε σε περισσότερη ευελιξία, ακόμη και στην μέγιστη δυνατή ευελιξία, ώστε να έχουμε κατάλληλες δεσμεύσεις πληρωμών, δεσμεύσεις πληρωμών, ε, πιστώσεις πληρωμών που να ικανοποιούν τους όρους των αντίστοιχων υποχρεώσεων. Όπως άλλωστε είχε ζητηθεί και από τους Προέδρους στην αρχή της συνεδριάσεως. Και υπογραμμίζω ότι η επισημάνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, διαδραμάτισαν ζωτικό ρόλο σε ολόκληρη τη διαδικασία, ίσω πολύ περισσότερο από ό,τι μπορεί να περιμένατε εσεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί το Κοινοβούλιο έχει υπογραμμίσει ότι οι δαπάνε Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν ευθέω να συγκριθούν με τι εθνικέ δαπάνε, γιατί επικεντρώνονται σε δυναμικό επενδυτικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατήρησε ζωντανό το ζήτημα των ιδίων πόρων, που ορισμένα κράτη-μέλη θεωρούσαν ότι είναι προτιμότερο να μην συζητηθεί, να μην εξεταστεί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με κάποια επιτυχία μπόρεσε να εισαγάγει μία ε, ρήτρα ευελιξίας αλλά και ρήτρα αναθεώρησης ε, αμφότερες δε καταγράφονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Επίσης υπογραμμίζει την ανάγκη να μετακυλιστούν οι πόροι στους νέους τομείς πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ότι αυτό μπορεί να μην ε, υλοποιείται στο βαθμό που το είχε ζητήσει με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκή Επιτροπή η αδίποτε σύγκριση με το, τα ίδια βλέπουμε όπως και πριν, η, ότι δηλαδή το τωρινό πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι το ίδιο με το προηγούμενο, νομίζω ότι καταρρύπτεται γιατί η αύξηση είναι σημαντική. Μπορεί στο συνολικό επίπεδο των δαπανών και θα υπογραμμίσω ότι είχαμε στη διαπραγμάτευση του προηγούμενο δημοσιονομικό πλαίσιο μείωση πολύ σημαντικότερη ω προ τι προτάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μείωση 13% στο προηγούμενο ποδοπού, ενώ τώρα έχουμε 8% μείωση. Και οι τελευταίε προτάσει δείχνουν ότι μπορούν οι ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδείξουν σημαντικό αίσθημα ευθύνη. Ωστόσο, και εμεί γνωρίζουμε και το περιμέναμε ότι θα μπορέσει να εξευρεθεί τελική λύση με το Κοινοβούλιο. Ήθελα να επενθυμίσω στους συναδέλφους ότι οτιδήποτε και να αποφασίσει οτιδήποτε αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τροποποιήθηκε Πράγμα το οποίο υποχρέωσε και το Συμβούλιο αλλά και την, την αναλασσόμενη Προεδρία να προβεί σε διάλογο και διαβουλεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ιδιαίτερα θα ήθελα να υπογραμμίσω την σημασία του άρθρου 15 τη συνθήκη, όπου αναφέρεται ο προσδιορισμό των γενικών πολιτικών επιλογών και κατευθύνσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση από πλευρά του Συμβουλίου. Τώρα, εμεί από πλευρά του Συμβουλίου καλούμε το Κοινοβούλιο σε διάλογο και διαπραγμάτευση για την ολοκλήρωση των απαραίτητων νομοθετικών πράξεων και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτό το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει από 1η Ιανουαρίου του 2014 να τεθεί ενισχύ και σε αυτό ε, στηρίζουν πολλέ ελπίδε οι δικαιούχοι. επίση, ένα πολύ σχημερός παράγοντα προβλέψιμότητα είναι απαραίτητο, διότι αν δεν, δεν έχουμε αυτό το παράγοντα προβλεψιμότητας που προσφέρει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, μόνο με ενιάφου προπολογισμού μπορούμε να λειτουργούμε, ω εκ τούτου επιχειρήσει, κυβερνήσει, τοπικέ αρχέ, δημοτικέ αρχέ, περιφερειακέ αρχέ ανά την Ευρώπη βρίσκονται σε πολύ μεγάλη δυσκολία και δεν θα μπορούν να αναπτύσσουν μακροπρόθεσμα σχέδια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όπου η εμπιστοσύνη στις οικονομίες μας αρχίζει δειλά-δειλά να επανέρχεται, η επταετής αυτή προοπτική ενός προϋπολογισμού για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα. Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε καθυστέρηση ή βραδιπορία, καλό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να ολοκληρώσουν ταχύτατα τι διαπραγματεύσει του και η ε, εναλλακτική, το να επανέλθουμε στενότατα επίπεδα και τα σε σχέση με το προηγούμενο και, και, και τις συνθήκες αντίστοιχες με αυτού του προηγούμενου πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου θα μας ε, κάνει να χάσουμε τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε επιτύχει και θα οδηγήσει σε αδέξοδο σε σχέση με την ισχύουσα νομική ε, βάση. Σας καλώ λοιπόν και εσάς και το ε, Συμβούλιο μέσω τη Ιρλανδική Προεδρία να προχωρήσετε στι διαπραγματεύσει για να συμφωνήσετε σε ένα πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο με ανοιχτέ συζητήσει στηριζόμενε σε πραγματικά στοιχεία και δεδομένα που είναι η μόνη πραγματική και ρεαλιστική λύση. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, πέραν του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου συζητήσαμε για τα ζητήματα του εμπορίου στην ε, διάσκεψη στη Σύνοδο αυτή, γιατί το εμπόριο μπορεί να προσφέρει πολλά και για την ανάπτυξη και τι εργασίε, αλλά και για επενδύσει δυνατέ και χάρη στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Με το πράσινο φως λοιπόν που δόθηκε για την ε, επανεκκίνηση, την ανεκκίνηση μάλλον διατλαντικών ε, συνομιλιών για εμπορικέ σχέσει, κατέληξε σε μια κοινή διακήρυξη του Προέδρου Ομπάμα, του υποφαινομένου και του Προέδρου Μπαρόσο και έτσι θα ξεκινήσουν οι εσωτερικέ διαδικασίε τώρα στα θεσμικά όργανα για να ξεκινήσουν διαδικασίε, διαπραγματεύσει για μια εταιρική σχέση εμπορίου και ε, συναλλαγών με τι ΗΠΑ. Παρακολουθούμε επίση εξελίξει στον αραβικό κόσμο δύο χρόνια μετά την έναρξη της Αραβικής Άνοιξης πρέπει να καταγραφεί και η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωξης στις ε, δημοκρατικές εξελίξεις της χώρες αυτές. Οι δε πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν πόσο ε, μεγάλα προβλήματα μπορούν να πορεύουν από αυτές τις εξελίξεις. Η Ευρώπη όμως παραμένει στρατευμένη και προσιλωμένη στο στόχο αυτό. Εν τέλει για το Μαλί ε, θα ήθελαμε να υπογραμμίσουμε ότι η αποφασιστική δράση πλευρά της Γαλλίας με την υποστήριξη και άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων και αφρικανικών κρατών έχει την πλήρη υποστήριξη Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία καταβάλει κατά δυνατή προσπάθεια και να τα απαραίτητα μέσα για την επαναφορά τη δημοκρατία και τη δημοκρατική τάξη και τη δραματική τάξη στο Μαλί. Ε, η Ευρωπαϊκή Αποστολή έχει βέβαια τεράστια σημασία στην υπόθεση αυτή. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, έτσι ολοκληρώνω την έκθεσή μου και καταγραφή των συμπερασμάτων και εργασιών του Συμβουλίου. Περιμένω τα σχόλιά σα. Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ. κύριε Πρόεδρε Δίνω τώρα το λόγο στον Πρόεδρο κύριο Μπαρόζο. Mr. President, Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, προκειμένου να συζητήσουμε τα αποτελέσματα της συνάντησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 7 και 8 Φεβρουαρίου. Πριν μπω στην ουσία, το νέο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο δηλαδή, επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που συζητήθηκε εκεί. Πρόκειται για το εμπόριο. Τα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν είναι πολύ σημαντικά. Ξέρετε ότι πριν από μερικέ μέρε ο πρόεδρο των ΗΠΑ, ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και εγώ ο ίδιο, ανακοινώσαμε την εκκίνηση μια διαδικασία που έχει ως στόχο να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ Ευρώπη και ΗΠΑ. Διατλαντική δηλαδή εμπορική συνεργασία. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ατζέντα μας υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ξέρετε, η ανάπτυξη και απασχόληση πόσο πολύ μα απασχόλησαν και στα πλαίσια των συζητήσεων για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Μια μέρα πριν το συμβούλιο αυτό στο Στρασβούργο θα θυμόσαστε ότι είχα πει ότι θέλουμε μια συμφωνία η οποία να αντικατοπτρίζει τις συμφωνίες που έχουμε κάνει μέχρι τώρα για την ανάπτυξη, την απασχόληση και του στόχου του 2020 ότι θέλαμε να ενισχύσουμε τη συνοχή, την κοινή γεωργική πολιτική, την εξωτερική πολιτική και να δείξουμε επίσης την αλληλεγγύη μας προς τους πιο αδύναμους. Ε, μίλησα επίσης υπέρ πιο ενισχυμένη ευρωπαϊκής διάστασης του προπολογισμού της Ευρώπης και της προστιθέμενης αξίας που δίνουν όλα αυτά. Στο Συμβούλιο υπενθύμησα στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων αυτά ακριβώς τα ίδια σημεία κάποιες κυβερνήσεις έκαναν τεράστιες προσπάθειες να πετύχουν μια συμφωνία που να τα καλύπτει όλα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι το επίπεδο της, του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου ήταν χαμηλότερο από αυτό που αρχικά είχαμε προτείνει. Με επιπλέον μειώσεις και με διαφορετική κατανομή ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες. Αυτή όμως είναι η πραγματικότητα μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης μεταξύ 27 χωρών μελών όταν απαιτείται ομοφωνία. Το επίπεδο λοιπόν των 960 της ε, πιστώσεων υποχρεώσεων και 908 πιστώσεων πληρωμών ήταν μια καλή πιστεύουμε ισορροπία στην οποία κατέληξαν τα κράτη-μέλη μετά από τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις διαπραγματεύσεις που ακολούθησαν κυρίως με τους καθορούς εισφορείς οι οποίοι ήθελαν μεγαλύτερες ακόμα περικοπές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φυσικά θα προτιμούσε ένα πιο φιλόδοξο σχέδιο. Είπα στο Συμβούλιο ότι τα επίπεδα που συμφώνησαν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είναι πιο κάτω από τις φιλοδοξίες που επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της ανάπτυξης και της απασχόλησης τα επόμενα χρόνια στην Ευρώπη. Τώρα, όσον αφορά την απόφαση στην οποία ομόφωνα κατέληξε η ενεργή κρατών και κυβερνήσεων, τώρα είναι η σειρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνεχίσει συζητήσει με το Συμβούλιο και θα είναι παρούσα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, παρά τις μειώσει αυτές πρέπει να αξιολογήσουμε με ισορροπία και αντικειμενικά το αποτέλεσμα να λάβουμε υπόψη μας δηλαδή ότι θέλουμε να στηρίξουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη. Συνεπώς, τα βασικά στοιχεία έχουν διατηρηθεί, όπως η διατήρηση της, ε, ε του προγράμματος ε, ε, συνδέοντας την Ευρώπη, Connecting Facility for Europe. Εκεί τα ποσά είναι παραπάνω από ό,τι έχουμε στην τρέχουσα περίοδο, όπως και τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Για τις μεταφορές επίσης υπάρχει μια αύξηση από τα 8,5 δις σε πάνω από 24 δις για την επόμενη περίοδο. Και για πρώτη φορά έχετε 5 δις για να επενδύσετε στις υποδομές για την ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε να αυξήσει επίσης σημαντικά τον προπολογισμό για την έρευνα και την καινοτομία και για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και για τον έρασμο για όλους. Για πρώτη φορά επίσης έχουμε ειδικό πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το πρόγραμμα COSME. Επίσης είναι πολύ σημαντικό ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να δημιουργήσει μια νέα πρωτοβουλία Κάτι το οποίο συζητήσαμε και στην τελευταία ολομέλεια μαζί. Με 6 δισεκατομμύρια ευρώ προπολογισμό, αυτό δείχνει μια δέσμευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε τις πολιτικές και κοινωνικές προκλήσεις που ε, αντιμετωπίζουν οι νέοι μας σήμερα στην Ευρώπη. Είναι η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης μας. Θέλουμε να χτίσουμε δηλαδή πάνω στην πρωτοβουλία που ξεκίνησαν 8 ε, χώρες πέρσι. Επίσης θα μας βοηθήσει σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο. Επίσης χαίρομαι πάρα πολύ που διατηρήσαμε και το πρόγραμμα βοήθειας για τους πιο αδύναμους. Υπήρχε βέβαια αντίθεση από ορισμένε πλευρέ. Παρ' αυτά πιστεύω ότι πετύχαμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ορισμένοι πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλεγαν ότι επειδή υπάρχει επικουρικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να βοηθάει τους πιο αδύναμους στις κοινωνίες μας. Ευτυχώς δεν κέρδισε αυτή η άποψη και χαίρομαι γι' αυτό. Τα ποσά τώρα που πάνε στη συνοχή και στη γεωργία είναι πολύ σημαντικά. Και πιστεύω ότι θα πετύχουν να βοηθήσουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Είναι μια δέσμευση που έχουμε αναλάβει για όλες μας τις πολιτικές, όπως επίσης το πρασίνισμα της γεωργίας μας, που είναι αξιοσημείωτο. Είναι μια δέσμευση που έχουμε υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Υιοθετήσαμε επίση ε, νέου κανόνε για τη συγχρηματοδότηση και την προχρηματοδότηση για να λάβουμε υπόψη μα τι ιδιαίτερε καταστάσει που επικρατούν στι πιο ευάλωτε χώρε μέλη. Χωρί τι διατάξει αυτέ, κάποιε χώρε ε, μέλη απλώ δεν θα ήταν σε θέση να κάνουν τι δημόσιε επενδύσει που θα έπρεπε να κάνουν τώρα, το 2014, το 2015. Χρειάζονται όμω τι επενδύσει αυτέ επιγόντω με τι διαπραγματεύσει και κατά τι διαπραγματεύσει εγώ επέμενα ότι δεν μπορεί να υπάρχει πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο χωρί την συμφωνία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι στόχοι ήταν σαφεί ήδη από την προσωρινή έκθεση που υιοθετήσατε εσεί τον Οκτώβριο και ο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του ε, ανέφερε ρητά κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου αυτού. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία λοιπόν ότι η Ιρλανδική Προεδρία Τώρα πρέπει να αρχίσει τις ε, διαδικασίες ε, συζητήσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το σημαντικό πάντως στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο είναι η ευελιξία, η ελαστικότητα, κάτι που κι εσείς έχετε ζητήσει. Γιατί πράγματι, όπως είπα και εγώ ίδιο στο Συμβούλιο, χωρίς αρκετή ελαστικότητα και ευελιξία, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, έτσι όπως έχει συμφωνηθεί, δεν θα μπορεί να δουλέψει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι η διαφορά του 51,5 δισεκατομμυρίων ευρώ ανάμεσα στις υποχρεώσεις και στις πληρωμές στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι κάτι που μπορεί να γίνει αποδεκτό εφόσον υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο ελαστικότητας για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό, μεταξύ άλλων, χρειαζόμαστε τη δυνατότητα να μπορούμε να μεταφέρουμε ε, ποσά που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί οι πληρωμές από τη μία χρονιά στην άλλη. Είναι ζωτική σημασία σε αυτό το σημείο. Δίνω μεγάλη σημασία στο θέμα της ελαστικότητας μεταξύ ετών και μεταξύ κατηγοριών για να καλυφθεί ακριβώς αυτή η διαφορά που έχουμε ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις πληρωμές. Και δεν πρόκειται μόνο για ένα τεχνικό ζήτημα, είναι θέμα ουσιαστικότατο. Γιατί την πραγματικότητα είναι τόσο σημαντικό όσο και τα συνολικά ποσά των πιστώσεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε αποτελεσματικά να δαπανίσουμε τα ποσά και τα κονδύλια που έχουν προβληθεί. Το πώ θα το καταφέρουμε αυτό θα εξαρτηθεί από τι λύσει που θα βρίσκουμε βάσει τη ελαστικότητα. Και όταν λέω ελαστικότητα, εννοώ την όσο γίνεται μεγαλύτερη ελαστικότητα. Πιστεύουμε επίση και εμεί ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων ε, όντως ε, βρίσκεται στο τραπέζι και πρέπει να εξεταστεί σοβαρά. Ε, ξέρω ότι εσεί θέλετε την επαναθεώρηση στα μέσα του δρόμου του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου. Εμείς ξέρουμε ότι είναι για 7 χρόνια, αλλά όντως στα μέσα του δρόμου θα πρέπει να επανεξαρθεί. Και αυτό το είπα και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπεύθυνη για τον προπολογισμό και πρέπει να διασφαλίσει ε, χρηστή ε, διαχείριση των κονδυλίων, των δαπανών και να τεθεί σε εφαρμογή η ελαστικότητα που θέλει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τέλο, επιτρέψτε μου να αναφερθώ λιγάκι στον προπολογισμό των φετινό και να σα πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τι ανησυχίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τα επίπεδα των πιστώσεων υποχρεώσεων. Η παρουσία των τριών θεσμικών οργάνων στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς υπεγράφει συμφωνία όπου προβλεπόταν ρητά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει επιπλέον πιστώσεις υποχρεώσεων εφόσον έχουμε την απόδειξη ότι ο εγκεκριμένο προπολογισμό δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες. Και να που έχουμε φτάσει ακριβώς σε αυτό το σημείο. Αυτό μπορούμε να το πούμε με σαφήνεια σήμερα. Προβλέπει επίσης η δήλωση αυτή ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα ε, αποφασίζουν όσο γίνεται πιο γρήγορα για οποιοδήποτε τροποποιητικό προπολογισμό για να αποφύγουμε ε, διακοπέ ή ελλείψεις ε, στι πληρωμέ και τι υποχρεώσεις. Αξιότιμοι ευρωβουλευτές, ξέρουμε ποιε είναι οι πρώτε πολιτικέ αντιδράσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην πολιτική συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι επικεφαλεί κρατών και κυβερνήσεων. Οι σημερινέ συζητήσει σίγουρα θα αποτελέσουν ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στην όλη διαδικασία προκειμένου να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Από εκεί και πέρα, εμείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παίξουμε τον δικό μας ρόλο προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατόν συμφωνία. Όχι μόνο για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, αλλά για τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι προσδοκούν από εμάς τα θεσμικά όργανα και τους εκλεγμένους τους καλά αποτελέσματα για τους ίδιους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Μπαρόζο. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Ντόλ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αγαπητέ κύριε Βαν κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητέ κύριε Μπαρόζο, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Η τελευταία σύνοδος κορυφής της Ένωσης, το μόνο που είχε ως ευρωπαϊκό ήταν το όνομα. Ήταν ένα ε, μια συνάντηση παζαριού κυρίως. Αποτέλεσμα έχουμε το χαμηλότερο ιστορικά προπολογισμό τη Ένωση. Ξέρω αγαπητοί φίλοι ότι πρέπει να το Υποστηρίξτε, Ξέρω, η ηρωνία είναι ότι τη στιγμή που οι αρμοδιότητες της Ένωσης αυξάνονται περισσότερο από ποτέ, σε μια φάση όπου πολλά κράτη δεν μπορούν να αντέξουν περισσότερο μόνα τους, οι πολίτες μας έχουν την ανάγκη της Ευρώπης θα προσέθετα ο υπολογισμό αυτό έτσι όπω έχει δεν είναι αποδεκτό. Υπενθυμίζω σε ορισμένα κράτη-μέλη ότι η κοινότητά μα θεσπίζεται στην αρχή της υπεροχής του δικαίου, μια συνθήκη που είναι το ανώτατο, ο νόμος. Το δημοσιονομικό πλαίσιο ωστόσο που μας προτείνεται αντιβαίνει στη συνθήκη. Πρώτον, διότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπερεύει τις αρμοδιότητές του παρακάμπτοντας την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Αυτό είναι μια παραβίωση του νομοθετικού ε, της του Κοινοβουλίου. Επιπλέον, προβλέποντας πιστώσει πληρωμών 50 δισεκατομμύρια χαμηλότερα από τι δεσμεύσει υποχρεώσεων, λέει, στην ουσία σημαίνει δημιουργία ελλείμματο. Ελλείμματο που είναι αντίθετο με του κανόνε που περιλαμβάνει η συνθήκη, που μα επιβάλλει την δημοσιονομική ισορροπία. Άλλωστε το 2012 ε, το δι, είδατε αυτό με μια ε, με ένα έλλειμμα 16 δισεκατομμύριων ευρώ η φιλοδοξία σας στα επόμενα έτη είναι να αναβάλλετε τις αποφάσεις, τις ουσιαστικές αποφάσεις στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Θα ήταν καταστροφή και θα έδειχνε ότι αυτό που γίνεται σε κράτη που είναι συνεχώς σε φάση πτώχευση αρχίζουν και γίνεται και στην Ευρώπη. Αυτά το είπατε κύριε Μπαρόζο, δεν αρκεί να το επαναλάβατε. Εμείς υπογράψαμε και τα τρία όργανα ότι δεν θα, υπάρχουν δεν θα υπάρχει έλλειμμα και τούτο πρέπει να γίνει σεβαστό και ανησυχώ από την εξέλιξη των γεγονότων. Η Ευρώπη μετά από μια τέτοια σύνοδο κορυφή πηγαίνει προ την κακή κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να υπεκφύγουμε τον αρμοδιο των ευθυνών μα. Έχω την εντύπωση μερικέ φορέ ότι η αλληλεγγύη απλά είναι μια λέξη. Και έχω δυστυχώ την θλιβερή εντύπωση ότι η βάση τη διαπραγμάτευση είναι η έκπτωση ή η αποτυχία μια ιδέα της Ευρώπης που παρασύρεται από την, ε, τους εθνικούς εγωισμούς. Εγώ δεν έχω αυτό το όραμα της Ευρώπης. Θέλω μια ισχυρή Ευρώπη που στηρίζεται στην κοινωτική μέθοδο και ομολογώ ότι έχω απογοητευτεί από πολλούς αρχηγούς κρατών κυβερνήσεων, όχι όλους, που έδειξαν ότι δεν βλέπουν μακριά και αγνόησαν την προστιθέμενη αξία της Ευρώπης. Είμαι απογοητευμένο επίση από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η νέα συνθήκη και είμαι υποχρεωμένο να το πω, αγαπητέ Πρόεδρε Αγαπητέ Ερμαν, μεταξύ των θεσμικών οργάνων δεν δουλέψαμε όπως έπρεπε να δουλεύουμε. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να προσεγγίσουμε τις απόψεις ε, τις δικές σας με το Κοινοβουλίο. Αυτό είναι μια διαπίστωση. Γνωρίζω επίσης ότι γνωρίζω επίσης ότι ουδέποτε έλαβε κάποιος υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου. Εμείς το είπαμε, το προειδοποίησαμε. Μα ζητάτε τώρα να είμαστε υπεύθυνοι. Αγαπητέ Πρόεδρε, ας καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι και ας είμαστε ανοιχτοί καταρχάς. Δώστε μας τις λεπτομέρειες της συμφωνίας της τελευταίας Συνόδου Κορυφής. και ας, ξε, ε, διαφωτίσουμε την εικόνα για τις ευρωπαϊκές πολιτικές, όχι μόνο με γενικούς τίτλους. Άλλαξε η Ευρώπη, κύριε Πρόεδρε, με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Το ξέρετε από τη θέση που είσαστε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα πιο ισορροπημένο σύστημα. Είμαστε συνομοθέτες, ισότιμοι συνομοθέτες. Τούτο ωστόσο δεν αφαιρεί ουδόλως το δικαίωμά μας να πούμε ναι ή όχι. Τα κράτη-μέλη τώρα μα έκαναν μία πρόταση Ας διαπραγματευτούμε και ας εφαρμόσουμε τη συνθήκη. Και πιστέψτε με, βάσει της συνθήκης θα είμαστε, θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Θα, αγαπητοί συνάδελφοι, ο προπολογισμό αυτός αποτελεί ένα μόνο το εκατό του ΑΕΠ. Είναι το ποσό πάνω στο οποίο δεσμευθήκαμε για ανακεφαλαιοποιήσουμε τις τράπεζες της Ισπανία. Είναι το ίμιση αυτού που δώσαμε στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τη δημοσιονομική κρίση. Είναι πολλά και είναι λίγα δεν μετράνε ωστόσο, δεν μετράει μόνο η ποσότητα, αλλά το νόημα που δίνουμε. Τα 27 κράτη δεσμεύθηκαν με 1% του ΑΕΠ τους για κοινέ πολιτικές, επεν, κοινέ επενδύσεις, για ένα κοινό μέλλον εν ολίγη. Αγαπητέ πρόεδρε Ρομπάη, έχουμε επίγνωση των ευθυνών μας. Μετά τις δηλώσεις σας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής σας διαβεβαιώνω ότι το Κοινοβούλιο δεν είναι μια συνέλευση παλαβών. Δεν ζητάμε τεράστια τεράστιο προπολογισμό. Ζητάμε έναν ρεαλιστικό προπολογισμό που προετοιμάζει το μέλλον και είναι δίκαιο μεταξύ των χρόνων. Ρεαλιστικό προπολογισμό που θα επιτρέψει να τιμήσουμε τι ευθύνε μα και ρεαλιστικό γιατί θα πρέπει να ενισχύσουμε τι κοινέ μα πολιτικέ που είναι πολιτικέ επενδύσεων. Ρεαλιστικό προπολογισμό τέλο γιατί ουδέποτε δεν πρέπει να είναι ελληματικό και θα εμείνουμε στη θέση στο ζήτημα αυτό, δεν θα προχωρήσουμε προ ένα έλλειμμα. Αυτό που θέλουμε, Πρόεδρε, είναι μια ε, ξεκάθαρη συμφωνία με ρήτρα να θεωρεί σε δύο ή τρία χρόνια να επανεξετάσουμε τον προπολογισμό. Δεν θα δεχθούμε ποτέ έναν προπολογισμό λιτότητα για 7 χρόνια. Δεν είναι σοβαρά τα πράγματα αυτά. Χρειάζεται λοιπόν τουλάχιστον η ρήτρα αναθεώρηση. Αυτό που ζητάμε είναι η εισαγωγή μια πραγματική ευελιξία. Ευελιξία μεταξύ 2011-12, 2012-2013 είχαμε αλλά είδατε τι σημαίνει ε, ευελιξία. Μας λείπουν 16 δις. Αυτό που χρειάζεται επίσης είναι αποτελεσματικότητα. Ζητάμε λοιπόν ίδιου πόρου, ώστε ο προπολογισμό της Ένωση να μην υπόκειται συστηματικά σε εκβιασμού. Δεν είναι παράλογε απαιτήσει μεταξύ μας, και αυτό είναι το αστείο, μεταξύ μας. Αν οι ευρωβουλευτές δεν έχουν το, την εξουσία να αναθεωρήσουν τον προπολογισμό τότε τι κάνουμε, γιατί κάνουμε εκλογές το 2014. Ας γλιτώσουμε τα λεφτά αυτά και ας τα κάνουμε, ας τις κάνουμε τις εκλογές το 2019. Εμείς παλεύουμε για την Ευρώπη, όχι για μια, ένα άθροισμα διακυβερνητικό. Παλεύουμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγει και υποστηρίζει κοινέ πολιτικέ για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Πιστεύουμε σε μια Ευρώπη που λαμβάνει σοβαρά τις δεσμεύσεις της, όπου το κράτος δικαίου είναι σεβαστό και πιστεύουμε ιδίως σε μια Ευρώπη που προστατεύει στους δύσκολους καιρούς από αυτή την αυστηρή κρίση, αυτή την σκληρή κρίση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το λόγο έχει ο Πρόεδρος κύριος Σβόμποντα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, <clears throat> το σημαντικότερο που είπατε σήματα, σήμερα είπατε ότι καταγράφεται στον προπολογισμό ένα χάσμα για το οποίο θα πρέπει να γίνονται πραγματεύσει. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω ξεκινώντα ότι δεν μιλάμε για λεπτομέρειε αλλά για βασικέ αρχέ. Μόνο έτσι μπορεί να εγκριθεί ο προπολογισμό αυτό. Όπω έχει όμω τώρα αυτή η πρόταση, δεν μπορούμε να την εγκρίνουμε και δεν πρόκειται να βρει επουδενή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Και μα ζητάτε να πιστέψουμε ότι σημειώνονται πολύ σημαντικέ αυξήσει, αλλά το συνολικό ποσό είναι λίγο χαμηλό. Πώς θα καταφέρατε αυτό το θαύμα, το συνολικό ποσό είναι χαμηλότερο από το προηγούμενο και γενικά παντού να παρουσιάζεται αυτή, δεν το έχουμε καταλάβει και προφανώς δεν το δεχόμαστε. Επίσης, μας λέτε ότι για την έρευνα και την ανάπτυξη θα έχουμε πολύ περισσότερα να αξιοποιήσουμε. Μακάρι. Μακάρι. Αλλά μεγάλες προτεραιότητες με μικρά ποσά πάλι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Και δεν θα κάνω συγκρίσεις του πριν και του μετά θα κάνω σύγκριση με το τι χρειαζόμαστε τώρα. Αυτή είναι η βάση, αυτή πρέπει να είναι και η βάση των προτάσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από εκεί ξεκινήσαμε και χαίρομαι για τον τρόπο με τον οποίο μα υπερασπίστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο πρόεδρο τη. Και θα, πρέπει να επανέλθουμε σε αυτά που πρότεινε η πρόταση τη Επιτροπή. Καταρχά, έχουμε να κάνουμε μία ύφεση. Δεν χρειάζεται κανεί να είναι δικό ε, τη κεντσιανή θεωρία για να πει ότι χρειάζεται όχι ένα μεγάλο προπολογισμό, ένα άλλο προπολογισμό χρειάζεται και εδώ έχει γίνει σημαντικό λάθος. Βεβαίω ε, γίνεται δεκτή η εγγύηση για την νεολαία που πάντοτε εμεί του σοσιαλιστέ ζητούσαμε. Αλλά με τα 6 δισεκατομμύρια θεωρείτε ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε ριζικέ αλλαγέ σε μια τόσο βαριά πληττόμενη από την ανεργία νεολαία τη Ευρώπη. Και μέσα στην τεράστια κοινωνική κρίση που αντιμετωπίζουμε, αρκούν αυτά τα ποσά και το κοινωνικό ταμείο. Δεν μου φαίνεται πιθανόν. Μιλήσατε για την παγκόσμια μας ευθύνη. Το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση, αντιμετώπιση των συνεπειών τη παγκοσμιοποίηση, γιατί έχει τόσο χαμηλή πρικοδότηση σε μια τόσο κρίσιμη εποχή για ολόκληρο τον κόσμο. Δεν δείχνει υπευθυνότητα αυτή τη Δεύτερον, ανταγωνιστικότητα. Όλοι μιλούν για ανταγωνιστικότητα, πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική η Ευρώπη, πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα τη Ευρώπη. Ε, αυτό δεν γίνεται όμω με τι μειώσει του μισθού και τι συντάξει. Βεβαίω χρειάζονται περισσότερε υποδομέ, βεβαίω προτείνεται κάτι τέτοιο, αλλά αλλά και μαζί με την ψηφιακή, ε, ψηφιακή ατζέντα και τις υποδομές για τις ε, ε, επικοινωνίες. Δεν βλέπω να αρκούν τα ποσά τα οποία προτείνει το Συμβούλιο ούτε καν για την εισαγωγή ενός συστήματος ευρυζωνικών ευρωζωνικού δικτύου και επικοινωνίων που θα μας φέρει στον 21ο αιώνα μπροστά. Και τρίτον, Ενισχύεται διαρκώ η φτώχεια σε όλη την Ευρώπη. Στην Νότια Ιταλία που επισκέφθηκα τι τελευταίε μέρε, βλέπω τι μπορεί να επιτευχθεί όταν διατίθενται αρκετά κονδύλια, αλλά μπορώ να δω επίση και να διαπιστώσω τι ακόμη λείπει. Οι προτάσει του Φαν και των αρχικών κρατών και κυβερνήσεων μα κάνουν να ντρεπόμαστε για αυτά που βλέπουμε να λαμβάνουν χώρα σε ορισμένε φτωχές περιοχέ τη Ευρώπη. Και εσεί, αν τι επισκεφτόσασταν, θα το βλέπατε αυτό. Ο κύριος Παρόσο μας λέει ότι μπορεί να δοθεί κάποια μικρή επιστηστική βοήθεια χωρί κανένα αποτέλεσμα. Αυτό είναι σκανδαλώδε το να λέτε ότι στην Ευρώπη δεν είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά τη φτώχεια. Αλλά υπάρχει μια ευρύτερη συζήτηση για τη μετανάστευση που μπορεί να προκαλεί η φτώχεια. Κυρίω από τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία. Αυτό απασχόλησε τη συζήτηση του Ηνωμένου Βασίλειου, τον κύριο Βαράζ, Φαράζ, ο οποίος ε, έκανε ε, τα παράπονά του για τη μετανάστευση από τη Βουλγαρία, προξενεί φτώχεια εκεί. Ναι, αλλά δεν βλέπω να λαμβάνονται πουθενά ουσιαστικά μέτρα. Ενισχύεται διαρκώ η φτώχεια και η μετανάστευση που αυτή προκαλεί. Βεβαίω, δεν έχετε άδικο σε αυτό. Ακόμα και στη Γερμανία έχει αυξηθεί ο αριθμό των φτωχών. Και καταλαβαίνω ότι κάποιο δήμαρχο μπορεί να πει πρέπει να δώσουμε αποφασιστικέ απαντήσει για να αντιμετωπίσουμε τις ροές των μεταναστών από τα κράτη-μέλη που προκαλεί φτώχεια. Αλλά όταν δεν υπάρχουν επαρκή κονδύλια για να στηριχθούν οι φτωχές περιοχές της Υπήρου μας, για να γίνουν επενδύσεις εκεί, για να μην υποχρεούται ο φτωχό εκεί να εγκαταλείψει την αιστεία του και να μεταναστεύσει κάπου αλλού, αλλά να έχει αρκετή βάση για να μείνει στη χώρα του και στην αιστεία του, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όσο και να διαμαρτυριόμαστε για τη φτώχεια και τη μετανάστευση που αυτή προξενεί στην Ευρώπη, χωρί να κάνουμε τίποτα όμω για του φτωχού, χωρί να κάνουμε τίποτα κατά τη φτώχεια, δεν φέρνουμε κανένα αποτέλεσμα. Και ένα τυπικό ζήτημα τώρα. Επτά ετία, επτά χρόνια. Μπορείτε κύριε Πρόεδρε εσείς να μου πείτε σε ποια χώρα καταρτίζεται επταετής προϋπολογισμός. Μακροπρόθεσμα έργα δεν έχει Βρετανία, δεν έχει Γαλλία, δεν έχει η Γερμανία με ενιαύσου προπολογισμού λειτουργούν τα κράτη αυτά, δεν έχουν επταετή προπολογισμού. Αυτή η επταετία λοιπόν είναι απαράδεκτη διάρκεια και θα ήταν παραδεκτή μόνο αν ήταν αρκετά μεγάλο ο προπολογισμό. Αλλά με έναν μήνυ προπολογισμό να μα λέτε ότι πρέπει να προγραμματίσουμε μια επταετία χωρί καμιά ελπίδα για ανάπτυξη στην Ευρώπη, τότε μιλάμε μόνο για μια επταετία λιτότητα στην Ευρώπη. Μιλάτε για μια ρήτρα αναθεώρησης. Ουσιαστική όμως ζητούσαμε εμείς, όχι μια επιφανειακή για τα φαινόμενα μόνο. Μια ρήτρα αναθεώρηση την οποία θα πρέπει να συμφωνήσουμε με την Ιρλανδική Προεδρία. Και αυτό βεβαίως επηρεάζει και την ευελιξία. Επισημάνατε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί περισσότερη ευελιξία και προσαρμογή στι νέε συνθήκε. Αυτά τα δύο απαραίτητα εκ των στοιχεία για τον προπολογισμό αυτό. Και για να ολοκληρώσω, δεν είναι το ζήτημα τα νούμερα. Το ζήτημα είναι η φιλοσοφία, η, η κοσμοθεωρία. Εάν θέλουμε να λειτουργήσει η Ευρώπη, τότε θα δώσουμε και τον σωστό προπολογισμό για να λειτουργήσει. Καταλαβαίνω ότι μπορεί ο κύριο Κάμερο να μην έχει όραμα την ε, προκοπή τη Ευρώπη. Αυτό που δεν καταλαβαίνω γιατί όλοι οι υπόλοιποι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τον ακολουθούν. Γι' αυτό λοιπόν εμεί όπω έχει αυτό ο προπολογισμό, για μα είναι απαράδεκτος, θα τον καταψηφίσουμε. Απαιτούμε ουσιαστικέ αλλαγέ στον προπολογισμό αυτό για να μπορέσουμε να τον δεχθούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σβόμποντα. το λόγο έχει ο κύριο Φεχόφστατ. Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να πω, κύριε Φανερομπάη, ότι η κριτική που θα ακούσετε από μένα δεν είναι προς το πρόσωπό σας, γιατί καταλαβαίνω πόσο πολύ δυσκολεύεστε να κάνετε 27 ηγέτες επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων να συμφωνήσουν μεταξύ τους και να καταλήξουν σε ομοφωνία. Τι να κάνουμε. Ο Τόνι Μπλερ το 2006 είχε πει ποτέ ξανά. Αλλά τελικά, να, που έχουμε το ίδιο και το ίδιο κάθε χρόνο. Η ανάλυση μου εμένα είναι ότι πρόκειται για copy-paste. Αντιγράφουμε το προηγούμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Έτσι είναι, με ελάχιστες διαφορές, όπως για παράδειγμα λίγο λιγότερα λεφτά στη γεωργία, λίγο περισσότερα στην καινοτομία, 27 στα 7 χρόνια, εκατομμύρια, κάτω από 5 εκατομμύρια το χρόνο για την έρευνα και την καινοτομία. Αυτό λέει ο προπολογισμό. Δηλαδή 4% του ετησίου προπολογισμού που πήγε από τη μία μεριά στην άλλη. Ενώ η Επιτροπή είχε ζητήσει το διπλό. Κατά τα άλλα, copy-paste του περσινού, της προηγούμενης μάλλον περίοδου του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου της προηγούμενης περίοδου. Το ίδιο με εξαιρέσει, με Τώρα 73 εξαιρέσει έχουμε, επιστροφές και τα έχω αυτά, έχω τον κατάλογο με όλα αυτά. Ναι, 41 είχαμε την προηγούμενη φορά, τώρα έχουμε 53 επιστροφές, εξαιρέσεις, earmarks κλπ. κλπ. Για τα κράτη-μέλη. Το ξέρω, το έχω συζητήσει και με το Λαμασούρ. Το ίδιο με την ε, προηγούμενη φορά και ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερες εξαιρέσεις. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι αυτό το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ένα πρόβλημα γιατί δημιουργεί τελικά ένα δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι εννοώ. Το πραγματικό έλλειμμα. Ξέρετε κύριε Φανερομπάου Ήμουνα στο Βέλγιο υπουργό. Ξέρετε ότι τη δεκαετία του 80 ήταν το Βέλγιο ο άρρωστο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί? Γιατί κάθε χρόνο είχαμε όλο και περισσότερα ποσά στις πιστώσεις υποχρεώσεων από ό,τι στις πληρωμές. Και τελικά στη δεκαετία του 80 καταλήξαμε να έχουμε το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα από όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε. Και τώρα το ίδιο κάνει και η Ευρώπη. Το rollover, οι, πλη... οι υποχρεώσεις δηλαδή που δεν καλύπτονται από τις πληρωμές ήταν 60 δισεκατομμύρια το 2000. 130 δισεκατομμύρια το 2006. Φέτος, τα τέλη της χρονιάς αυτής, θα είναι 230 ή 250 ε, δις από ποσά που δεν καλύπτονται από πληρωμές και με τις νέες δημοσιονομικές ε, προοπτικές το πραγματικό έλλειμμα της Ευρώπης θα είναι πάνω από 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Οπότε τελικά δεν κλείνουμε το χάσμα, δεν γεφυρώνουμε τις διαφορές, αντίθετα τις κάνουμε ακόμα μεγαλύτερες. Και για να σας δώσω και τη σχέση ανάμεσα στις υποχρεώσεις και τις πληρωμές ήταν 95 την ε, προηγούμενη φορά και τώρα είναι 94. Ενώ θα έπρεπε να ήταν το αντίθετο. Θα έπρεπε να έχει αυξηθεί περισσότερο και να ήταν 100% αν δεν θέλουμε να έχουμε επιπλέον έλλειμμα. Συνεπώς, επίσημα, ενώ δεν πρέπει να έχουμε ούτε χρέος ούτε έλλειμμα, με αυτά τα ποσά θα έχουμε 300 δισεκατομμύρια ευρώ έλλειμμα δηλαδή που δεν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε. Ήδη πόρη τώρα. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι έγινε, γιατί η Επιτροπή είχε μια πολύ καλή πρόταση. Εκεί, κύριε Φανουροπά, εσείς την είχατε δεχτεί το Νοέμβριο. Το δεχτήκατε για τον ΦΠΑ από 1η Ιανουαρίου του 2021 και δεύτερον τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Οπότε θα μπορούσαν να ήταν πιο μικρά τα ποσά από τις διάφορες χώρες μέλη. Και τώρα, τίποτα. Ναι, θα δουλέψουν παραπάνω με το ΦΠΑ, θα σκεφτούν το θέμα των χρηματοπιστωτικών, του φόρου δηλαδή χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, αλλά τίποτα συγκεκριμένο. Καμία πρόταση. Και γι' αυτό είμαστε απογοτευμένοι, Πρόεδρε. Δεν πρόκειται για ένα δημοσιονομικό πολιτές πλαίσιο που να μπορεί να δεχτεί το Κοινοβούλιο και μία δυνατότητα μόνο υπάρχει ίσως να έχουμε μία ρήτρα sunset, δηλαδή προδευτικής ε, κατάργησης, ώστε μετά τις επόμενες εκλογές το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να πρέπει να εγκρίνει εκ νέου τις ε, προτάσεις αυτές, αν θέλουμε να τεθούν σε εφαρμογή. Είναι ο μόνος τρόπος ώστε δημοκρατικά να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε η κυρία Ντουιράν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν μας ε, προτείνουν προϋπολογισμό, αλλά μια, ε, ε, ένα πλεχτό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ένα κέντημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τις δαντέλες, με όλα. Τα πάντα είναι, προϋπολογισμός δεν είναι. Μιλήσατε για το τωρινό και το προηγούμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο κύριε Πρόεδρε, αλλά το συγκρίνεται με το προηγούμενο. Αυτό είναι λάθος. Ο προπολογισμό προετοιμάζει το μέλλον. Πώς το συγκρίνεται με κάτι του παρελθόντος 7 ετών πριν. Δεν είναι κάτι τέτοιο αν θέλετε να προωθήσουμε τις ε, αξιολογήσεις. Ο προπολογισμό αυτός δεν είναι καλός ούτε από το περιεχόμενο ούτε από τη μέθοδο. Έγινε χωρίς διαφάνεια. Ευχαριστώ τον κύριο Λαμασούρ ο οποίος τόνισε την ανάγκη να δούμε τα νούμερα. Δεν έχουμε τα νούμερα. Εμείς εκπροσωπούμε τους πολίτες, δεν έχουμε τα νούμερα. Προτείνω λοιπόν πέραν τη συζήτηση που θα κάνουμε να πούμε σαφώς με έναν, μπορούμε να δουλέψουμε με έναν προπολογισμό για το 2003 και 2014 και το 2014 να κάνουμε πραγματικές συζητήσεις εν ώψη των ευρωεκλογών, αφήνοντας τους πολίτες να κρίνουν αυτά, ούτως ώστε να δεσμεύσουν και το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Κάποια στοιχεία ωστόσο για τον προϋπολογισμό. Περικοπές. 90 δις σε 7 χρόνια. Κάμποσα. 12 δις για το 2013 και το 14 είναι σαφές ότι το θέμα της απόκλησης μεταξύ πληρωμών και υποχρεώσεων αναφέρθηκε. Δεν θα σας ε, εξηγήσω κύριε Βάνο Ρομπάη ότι αυτό είναι χιονοστιβάρα, το ξέρετε. Μπαίνουμε, οι αποκλήσεις μεταξύ πληρωμών και υποχρεώσεων μας βάζουν σε ένα σε μια λογική ελληματική που θα οδηγήσει τους πολίτες να πληρώσουν πολλά αυτά που δεν κάνουν οι κυβερνήσεις και που μας εμποδίζουν να έρθουμε να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη. Αυτό κάνουμε με τον προϋπολογισμό. Τρίτον, το θέμα των ιδίων πόρων. Μηδέν συμφωνία στου ίδιου πόρου. Πραγματικά λυπάμαι. Η μόνη φράση που βρήκατε είναι το could be θα μπορούσε. Συμφωνία είναι αυτή. Και για τον ΦΠΑ, ιδίω δε για τον φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Εδώ έχουμε ξεφύγει τελείω από αυτά που έπρεπε να είχαμε κάνει. Επικυρώνουμε στην ουσία μια σειρά ε, επιταγών για τους Βρετανούς και όχι μόνο για τους Ολλανδούς ε, για τους Αυστριακούς, για τους Γερμανούς, προσθέτουμε κι άλλο και για τους Δανού. Μέσα σε μια λογική κοινοτική τι ρόλα έχουν τα τσεκ και κάποια στοιχεία ευελιξία μας δίνουν και μια ρήτρα επανεξέταση Εξηγήστε μου πώς σε μια ρήτρα επανεξέταση σε δύο χρόνια το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ομόφωνα θα μπορέσει να κάνει αυτό που δεν μπορέσει να κάνει πριν από λίγε εβδομάδε. Εγώ δεν το καταλαβαίνω και δεν μπορώ να καταλάβω Καταλαβαίνω ποια είναι η κατάσταση, αλλά γιατί θα είναι σε καλύτερη κατάσταση σε δύο χρόνια για να αλλάξουν τον προπολογισμό ομόφωνα, ομόφωνα. Σίγουρα η ρήτρα επανεξέταση δεν είναι το εργαλείο που επιτρέπει να έχουμε μια καλύτερη συμφωνία για το θέμα του προπολογισμού. Δεν είμαστε τελείω καθόλου παράλογοι. Είμαστε λίγο πιο φιλόδοξοι, πιο τολμηροί, αλλά δεν είμαστε παράλογοι. Ε, δεν έχουμε από τη μια μεριά ένα συμβούλιο φρόνιμο και ένα κοινοβούλιο που παραλογίζεται. Θέλουμε έναν προπολογισμό που επιτρέπει επενδύσεις στην έρευνα, στην ανάπτυξη και τα ταμεία συνοχής που, και το ταμείο συνοχής που αναφέρεται προηγουμένως. Είναι εργαλεία συνοχής, είναι εργαλεία ανάπτυξης μέσα σε μια φάση κρίσης. Ε, είναι δεν μπορεί να συγκρίνουμε τις δυνατότητες που μπορούμε να δώσουμε με αυτό που μας δώσατε. Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να δεχθούμε, σίγουρα δεν μπορούμε να δεχθούμε το, το κείμενο αυτό, ίσως να το διαπραγματευτούμε, αλλά η μικρή πόρτα ανοιχτή που είδαμε μέσω της πρωτοπροτάσεών σας είναι ανεπαρκέστατη. Εγώ προτείνω μέχρι το 2014 και από το 2014 και μετά ας δουλέψουμε με βάση έναν ετήσιο προπολογισμό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τύραν. Ο κύριος αν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρόεδρε Φανερομπά, εκ μέρου τη ομάδα μου θέλω να σα ευχαριστήσω πολύ για, την, ε, για το έργο σα προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Δεν λέω ότι είναι τέλεια. Πιστεύουμε όμως ότι διέπεται από πραγματισμό και ισορροπία. Υπάρχουν χώρες που θέλουν περισσότερες δαπάνες και άλλες που θέλουν να προστατεύσουν τη δικιά τους θέση. Θα μπορούσαμε βέβαια να έχουμε μεταρρυθμίσει τον ε, ευρωπαϊκό προπολογισμό. Συμφωνώ με τι παρατηρήσει που έκαναν ε, άλλοι. Είναι μια προτεραιότητα όμω παρά τη ρητορική του κύριου Σόβοντα κλπ. Κατ' εικόνα του Πρόεδρου Ολάντ, εμείς πιστεύουμε ότι η προοπτική μας και η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να μειώνουμε τις διαφορές. Εμείς πιστεύουμε ότι περισσότερα χρήματα πρέπει να πηγαίνουν στην ανταγωνιστικότητα. Ο κύριος Ολάντ ε, ε, πρέπει να δει ότι το 40% του προπολογισμού μας εξακολουθεί να πηγαίνει στη Γεωργία, τώρα που είμαστε στον 21ο αιώνα. Τέλος πάντων, δεν ε, με εκπλήσουν βέβαια αυτά που ακούσαμε από τους επικεφαλεί των άλλων πολιτικών ομάδων, πάντως μην ξεχνάμε ότι τελικά είναι εθνικέ κυβερνήσεις και όχι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ε, κανονίζουν και βρίσκουν τα χρήματα για τις, ε, τους ίδιους πόρους. Εκείνοι που τα παίρνουν από τους ε, πολίτε, οι οποίοι πληρώνουν ΦΠΑ κλπ. από τα νοικοκυριά κλπ. οι οποίοι στην Ήπειρό μας τελικά συνεισφέρουν αυτόν τον τρόπο στους ιδίους πόρους. Οι ηγέτες από όλες τις μεγάλες ομάδες εδώ πιέζουν για αύξηση του προπολογισμού. Ο κύριος Κάμερον έχει πολλούς φίλους εδώ. Ο κύριος Ρίτε από τους Φιλελεύθερους, η κυρία Μέρκελ ε, από το ΕΛΚΑ. Αλλά ακόμα και από τους σοσιαλιστές κάποιοι, ναι, μιλάνε υπέρ της αύξησης αυτής. Την προηγούμενη εβδομάδα πήρα ένα email, πολλά πήρα δηλαδή, αλλά να, ήταν ένα το οποίο πρόσεξα ιδιαίτερα. Από ένα νέο από το ΕΛΚ. Από την νεολαία του ΕΛΚ. Λέει ότι η συμφωνία μετά από πολλούς μήνες διαπραγματεύσεων καταλήγει σε μια καλή ισορροπία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει υπεύθυνα να ψηφίσει για τη λιτότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιμένω, έτσι, νεολαία του ΕΛΚ. Μου το έγραψε αυτό. Τώρα θα έρθω σε αυτά που ακούσαμε για ελληματικό προϋπολογισμό. Η ερώτησή μου είναι απλή και είναι εξή. Οι άλλοι προπολογισμοί που έχουμε εγκρίνει δεν ήταν το ίδιο. Μην λέμε αυτά τα πράγματα. Ξέρουμε τελικά ποιο παιχνίδι παίζεται. Και κάτι το οποίο δεν αναφέρατε εδώ, αλλά το ανέφερε στην ομιλία του κύριο Σούλτς. Το θέμα της μυστικής ψηφοφορίας. Να θα είναι γελίο για το Κοινοβούλιο. Εμείς πρέπει να λογοδοτούμε στο εκλογικό μας σώμα και να είναι γνωστό το πώς ψηφίζουμε. Είναι μια από τις πιο σημαντικές ψηφοφορίες. Πρέπει να είμαστε σε θέση να δικαιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ψηφίζουμε. Συνεπώς, Πρόεδρε, δεν είναι μια τέλεια συμφωνία. Αλλά το κοινοβούλιο μας πρέπει να δείξει ότι μπορεί να σκίσει τις νέες του εξουσίες υπεύθυνα. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να τον στηρίξει. Αν αποφασίσει πόλεμο με το Συμβούλιο το κοινοβούλιο μας, είναι κάτι από το οποίο έχουμε όλοι να χάσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κανανάν. Ο Νούτελ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, θα πρέπει να ομολογήσω ότι αισθάνθηκα μια ευχάριστα, ευχάριστη έκπληξη όταν ένα Σάββατο πρωί άνοιξα τη τηλεόραση για να ενημερωθώ από τα πρωινά δελτία ότι αρχίζουν να βρίσκουν σωστές λύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Και είπα, Θεέ μου, Θεέ μου, αυτή την πικρία χειμωνιάτικη μέρα, μήπως τελικά είδαν την κοινή λογική οι Ευρωπαίοι ηγέτες, μήπως τελικά τους, ε, τους ε, συνέτησε ο Κάμερον και, ρώτη, και αναρωτήθηκα πού είναι το ψητό. Και ανακάλυψε το ψητό δεν ήταν μοσχαράκι. Το ψητό ήταν κρέας αλόγου. Αυτό δηλαδή ήταν ότι η νίκη του Κάμερον ήταν μια, ένα πουκάμισο αδιανό. Φαίνεται ότι τελικά ε, αυτές οι περικοπές είναι ελάχιστες και στην πραγματικότητα ο Βρετανός φορολογούμενος θα πληρώσει πιο πολλά τώρα, διότι θα αυξάνεται ε, το χρόνο και κάθε χρόνο η δική μας εισφορά στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Μπορεί να φαίνεται λοιπόν ως νίκη για τον Κάμερον αυτό το αποτέλεσμα, αλλά τελικά δεν μειώνεται η συνεισφορά μας. 53 εκατομμύρια λίρες πληρώνουμε για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό, ούτε μία δεκάρα παραπάνω το σκοπεύουμε να δώσουμε. Και τώρα βλέπουμε ότι η ομάδε στο κοινοβούλιο ζητούν μυστική ψηφοφορία. Και να σα ρωτήσω, τι φοβάστε, φοβάστε τα εθνικά σα κοινοβούλια, τα κοινοβούλια στι πατρίδε σα, ή μήπω τελικά πιο πολύ φοβάστε αυτού που σα εξέλεξαν και σα έφεραν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το να ζητηθεί μυστική ψηφοφορία για ένα θέμα τέτοια σημασία που ε, έχει να κάνει με τι συνδυσιακέ σα επιλογέ σε μια επιλογή, σε μια κρίσιμη εποχή λιτότητα και κρίση, ουσιαστικά σα μετατρέπει σε εκπροσώπου μια μπανανία και όχι σε σοβαρούς ευρωβουλευτές όπως θα έπρεπε να είστε. Ερωτώ λοιπόν και λέγω ότι δεν μπορεί να είναι τυχαίο πως η Financial Times σήμερα μια δημοσκόπηση που δημοσιεύουν αποδεικνύει ότι το 50% και άνω των Βρετανών προτιμούν να αποχωρήσει η χώρα τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να σας πω ευχαριστώ, ευχαριστώ που μας δείξατε και το δρόμο της εξόδου, μας ανοίξατε την πόρτα για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ η κυρία Λιωτάρη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Χαίρομαι που βρισκόμαστε εδώ για να ανταλλάξουμε απόψεις μεταξύ μας. Ζητάμε από τα κράτη-μέλη λιτότητα αυτό έχει νόημα εφόσον και εμείς στην Ευρώπη μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα. Τα δισεκατομμύρια έτσι κι αλλιώς που ξοδεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα πληρώνει ο Ευρωπαίος πολίτης. Η πρόταση που έχουμε μπροστά μας δεν πιστεύω ότι έχει τη σωστή κατανομή και αφήνει στο περιθώριο πολλές κοινωνικές ομάδες. Δεν ενισχύονται οι πιο αδύναμοι. Κύριε Φανερομπάου, πολύ ωραία τα λέτε. Τελικά όμως, διάφορα προγράμματα όπως είναι το ΙΤΕΡ, ο Γαλιλαίος, το ΤΣΙΕΣ κλπ. Τα βάζετε σαν προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης. Μα σε περίοδο κρίσης τα χρήματα πρέπει να πηγαίνουν απευθείας στους πολίτες. Με τέτοια ακριβά προγράμματα κύρους δεν ε, ενισχύουμε την κοινωνική ανάπτυξη. Ούτε τους νέους, ούτε τους μικρούς επιχειρηματίες. Όλοι αυτοί είναι δυνατόν να έρθουν ε, και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το Γαλιλαίο και άλλα τέτοια μεγάλα προγράμματα. Οι νέοι για να βρούνε δουλειά πώς θα το κάνουν, πώς θα ανταγωνιστούν τα άλλα προγράμματα που βάζετε εσείς μαζί στην ίδια κατηγορία. γίνονται περικοπές στα κοινωνικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ενισχύονται οι πιο αδύναμοι. Αντίθετα, είναι οι χαμένοι του νέου αυτού σχεδίου. Για μας η κοινωνική Ευρώπη είναι το πιο σημαντικό. Δυστυχώς δεν αντικατοπτρίζεται αυτό στην πρότασή σας. Οι πιο αδύναμοι και οι νέοι που ψάχνουν δουλειά, σύμφωνα με το δικό σας ε, πρόγραμμα, τη δικιά σας πρόταση, είναι οι χαμένοι της Ευρώπης. Το ίδιο θα έλεγα και για το κλίμα. Το περιβάλλον, τα σχέδια για την αλία θα πληρωθούν από τέτοια χρήματα που πληρώνουμε και την ε, γεωργία με τις ίδιες επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις όμως πηγαίνουν για την αύξηση της παραγωγής και για την εντατική γεωργία. Αλλά αυτό ζημιώνει το περιβάλλον, δεν το προστατεύει. Αντίθετα, οι μικροί αγρότες, οι πιο δύναμοι, βλέπουν τα χρήματα να περνάνε κάτω από τη μύτη τους χωρίς να μπορούν να υποφεληθούν καθόλου. Και δεν προστατεύεται το περιβάλλον. Για τη δικιά μας ομάδα είναι απαράδεκτο να βάζουμε το περιβάλλον σε δεύτερη μοίρα. Θέλουμε οικονομικές εγγυήσεις για το περιβάλλον. Αλλιώς δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε μια τέτοια πρόταση. Οι περικοπές στον προπολογισμό δεν λέω ότι είναι απαραίτητα κάτι αρνητικό, αλλά η πρόταση αυτή δεν είναι υπέρ ενό πράσινου προπολογισμού και αυτό είναι με το οποίο δεν συμφωνεί η ομάδα μας. Δεν θέλουμε περισσότερα χρήματα, αλλά θέλουμε καλύτερη κατανομή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λιωτά. Ο Στάσεν έχει το λόγο. Η κυρία Στάσεν. Ευχαριστώ πολύ. Ας ξεκινήσουμε με κάτι θετικό για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει πάντα περισσότερα χρήματα. Ποτέ δεν έχει αρκετά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη φορά δεν εξυπηρετείται. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ μικρό θετικό στην συμφωνία στην οποία έχουμε καταλήξει και έχουμε μπροστά μας. Και αυτό είναι ο, οι μειώσεις στον προπολογισμό αλλά είναι κάπως αποξηρωμένος. Η συνοχή που θέλουμε να είναι πιο αποτελεσματική μένει ανέπαφη. Σε άλλες πολιτικές ε, βλέπουμε να παραμένουν τα ίδια πράγματα. Οι μισθοί βλέπουμε ότι περικόπτονται. Και τελικά με το Στρασβούργο, πάμε στο Στρασβούργο το οποίο τόσο πολύ ζημιώνει το περιβάλλον. Οπότε γιατί να χαρούμε για αυτή τη συμφωνία. Ούτε και η Ολλανδία χαίρεται για αυτή τη συμφωνία διότι βάζετε εδώ προϋποθέσεις για την οικονομική ανάπτυξη. Δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τι λέει τώρα ότι θέλει να μπλοκάρει τη συμφωνία αυτή. Όχι όμω γιατί ξοδεύουμε όλο και περισσότερα. Όχι. Ο λόγο για τον οποίο θέλει να μπλοκάρει τον προπολογισμό αυτό είναι γιατί πιστεύει ότι δεν ε, υπάρχουν επαρκή κονδύλια. Δηλαδή να σπαταλάμε ακόμα περισσότερο. Οι μεγάλες ομάδες σπαταλούν τα χρήματα. Δεν συμφωνεί η δικιά μας η ομάδα, ούτε το δικό μας το κόμμα, με αυτά που κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα στην Ολλανδία. Είναι θλιβερό να βλέπουμε αυτά που λέει ο κ. Φερχόσταθ και ο κύριος Σούλτς, που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η υποστήριξη της δημοκρατίας, αλλά συγχρόνως ζητούν εδώ μυστική ψηφοφορία. Τι διαφάνεια είναι αυτή. Άρα δεν υπάρχει διαφάνεια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ναι, να ψηφίσουμε μυστική ψηφοφορία για να μην μάθει ποτέ ο Ευρωπαίος πολίτης τι αποφασίζεται κάτω από τη μύτη του και χωρίς να λογοδοτούμε σε αυτόν. Ευχαριστώ κύριε Στάσεν. Το λόγο έχει τώρα ο πρόεδρος κύριος Μπαρόζο. Δεν υπήρχαν απευθείας ερωτήσεις που τέθηκαν προς εμένα διότι αυτή είναι συμφωνία αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων όπου δεν ψηφίζει η Επιτροπή. Θα ήθελα ωστόσο με την ευκαιρία αυτή να σας πω τα εξή. Πρώτον, συμμερίζομαι τις ανησυχίες που εξέφρασαν οι περισσότεροι επικεφαλείς των ομάδων. Το ερώτημα είναι από εδώ και πέρα που πάμε. Τι κάνουμε μετά. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα πολιετέ πλαίσιο. Ξέρω ότι κάποιοι από εσά πιστεύουν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με άλλο τρόπο, σε αιτήσια βάση. Δεν συμφωνώ. Και σας λέω γιατί δεν συμφωνώ. Διότι κάποιες από τις περιφέρειες και χώρες που είναι οι πιο ευάλωτες χρειάζονται επενδύσεις τώρα. Η αναβολή θα ήταν λάθος. Και αν δεν υπάρχει πραγματικό ΠΔΠ. Δεν νομίζω ότι μπορούμε πραγματικά να συμφωνήσουμε έγκαιρα για τη νομική βάση που χρειάζεται για να επενδύσουμε, να δαπανίσουμε χρήματα που θα ξεκινούν από την 1η Ιανουαρίου του 2014. Αυτό που η έκκλησή μου λοιπόν προς εσάς και προς το Συμβούλιο είναι να ξεκινήσετε σοβαρές διαπραγματεύσεις για να πετύχετε ένα αποτέλεσμα για την Ευρώπη. Έχοντας βεβαίως υπόψη τις αρχές της ευρωπαϊκής ευθύνης. Στις αρχικές παρατηρήσεις μου μάλιστα ήδη έκανα ένα σχόλιο για την κατεύθυνση προς την να πρέπει να πάνε οι σοβαρές διαπραγματεύσεις, ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Η συζήτηση με σωστό τρόπο του θέμα της ευελιξίας. Επαναλαμβάνω αυτά που είπα στις αρχικές παρατηρήσεις μου. Και αυτό που είπα και στο ίδιο το Συμβούλιο χωρίς σωστά επίπεδα ευελιξία, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο όπως συμφωνήθηκε μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, απλά δεν θα μπορεί να λειτουργήσει. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η διαφορά 51,5 δις ευρώ μεταξύ των υποχρεώσεων και των πληρωμών στο επόμενο ΠΔΠ μπορεί να γίνει δεκτό μόνο στο μέτρο που έχουμε ευέλιξία συγκεκριμένη και μέγιστη για να μπορέσουμε να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις βάσει της συνθήκης. Ιδίως το άρθρο, βάσει του άρθρου 323. Για τούτο χρειαζόμαστε μεταξύ των άλλων προϋποθέσεων τη δυνατότητα να μεταφέρουμε ε, μη χρησιμοποιημένα περιθώρια κάτω από τα νοτορία από το ένα χρόνο στον άλλο. Αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Και είναι πολύ σημαντικό όταν μπαίνουμε σε διαπραγματεύσει, όταν μπείτε εσεί στι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο, Βεβαίω και η Επιτροπή είναι έτοιμη να βοηθήσει, πρέπει να δείτε όχι μόνο τα επίπεδα των πληρωμών, δηλαδή τα ανώτατα επίπεδα, αλλά και το τι πραγματικά δαπανάτε χρόνο με το χρόνο στον ετήσιο προπολογισμό κατά τη διάρκεια της, της περίοδου του ΠΔΠ. Αν συγκρίνουμε το, την κατάσταση των, του, του υφιστάμενου, της υφιστάμενης περίοδου ΠΔΠ, ε, Ιδίω τα έξι πρώτα χρόνια, δεν μπορώ να σα μιλήσω για το 13 ακόμα, γιατί ακόμα βρισκόμαστε στη φάση υλοποίηση. Αν κάνουμε πάντω τη σύγκριση πληρωμών και υποχρεώσεων τα τελευταία έξι χρόνια, διαπιστώνουμε ότι κατά κάθε χρόνο δαπανίσαμε κατά μέσο όρο 122,2 δις σε πληρωμές. Πραγματικές πληρωμές. Δεν μιλάω ούτε για υποχρεώσεις ούτε για νοτατόρια πληρωμών. Για πραγματικές πληρωμές κατά μέσο όρο. Για, το επόμενο, για την επόμενη περίοδο ΠΔΠ με συνολικό ανώτατο όριο πληρωμών στα 908,4 δις, ο μέσος όρος πληρωμών μπορεί να φτάσει τα 129,7 δις. Δηλαδή, 7,5 δις περισσότερο σε πληρωμές κάθε χρόνο για 7 χρόνια. Βεβαίως όλα εξαρτώνται, τέλος όχι όλα, τα περισσότερα εξαρτώνται από την σωστή λύση της ευελιξίας. Ευελιξία μεταξύ κατηγοριών, μεταξύ ετών, διότι όπως ξέρετε αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο είναι πολλοί πόροι να επιστρέφουν στα κράτη-μέλη διότι δεν χρησιμοποιήθηκαν, δεν αναλώθηκαν. Αυτό είναι η πραγματικότητα που έχουμε σήμερα. Ιδίω λόγω της έλλειψης απορρόφησης από πολλά κράτη-μέλη, μερικά από τα οποία έχουν εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο απορρόφησης. Πιστεύω ότι είναι δυνατό, αν υπάρχει καλή βούληση και από τις δύο πλευρές, να βρούμε μια λύση που θα μας επιτρέπει να πετύχουμε εν τέλει ένα συμβιβασμό. Γι' αυτό είπα σαφώς ότι έτσι όπως είναι δεν θα δουλέψει. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ ξεκάθαρη δήλωση. Και το λέω ενώπιόν σα, διότι είπα ακριβώ τα ίδια και δήλωση τα πρακτικά έκανα κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου. Με το σωστό επίπεδο ευελιξία, ωστόσο, όχι μόνο η μεταφορά μεταξύ ετών, τη μεταφορά μεταξύ ετών, αλλά και το αποθεματικό επίδοσης που συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ο κανόνας νη συν τρία που επιτρέπει στα κράτη που δεν μπορούν να δαπανίσουν σε δύο χρόνια τις ε, υποχρεώσεις τους αλλά να έχουν και ένα έξτρα έτος για να το κάνουν αυτό και με τη δυνατότητα να περνάμε από κατηγορία σε κατηγορία μπορούμε να βρούμε ένα δρόμο προς το μέλλον. Δεν λέω ότι θα είναι εύκολο, πιστεύω ότι θα είναι μια δύσκολη διαπραγμάτευση, είμαι βέβαιος συζήτησε το θέμα αυτό βέβαια όχι μόνο με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου αλλά και με τον, την Προεδρία του Συμβουλίου, τον Πρωθυπουργό Κένα από την Ιρλανδία και είμαι βέβαιος ότι αν υπάρξει βούληση στο τέλος θα βρούμε κάποιο συμβασμό. Διότι ο προπολογισμό αυτός, μάλλον ο, ο το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο αυτό είναι κρίσιμο για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη στην Ευρώπη και για την αλληλεγγύη που χρειάζονται ιδίω οι πιο τρωτέ περιοχές μας. Διότι σε ορισμένε περιοχές της Ευρώπης υπάρχουν κατάσταση πραγματικά κοινωνικού πανικού. Και αυτό που σας λέω είναι η δήλωση που έκανα και προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πιστεύω ακόμα ότι είναι δυνατό να επέλθει η συμφωνία αν υπάρχει το αναγκαίο πνεύμα μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Βαν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι καλό θα ήταν να μην ξεκινήσουμε μια ψευδεπίραπτη συζήτηση. Μια συζήτηση δηλαδή πάνω σε λάθο βάση, συζήτηση μεταξύ καλών και κακών Ευρωπαίων όπου οι κακοί Ευρωπαίοι είναι οι αρχή κρατών και κυβερνήσεων, χωρί να θέλω να διευκρινίσω ποιοι υποτίθεται ότι είναι οι καλοί Ευρωπαίοι. Εγώ όμω το αυτό μου το θεωρώ σκαλό καλό Ευρωπαίοι, Ευρωπαίο και α μην ξεκινήσουμε αυτή την ψευδεπηρεάτη συζήτηση, γιατί δεν είναι συζήτηση μεταξύ υπεύθυνων και μη και ανεύθυνων, όπως φάνηκε κάποιοι να λένε, δεν είναι σωστό αυτό δεν θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανήκει σε ένα στρατόπεδο. Βεβαίω είναι συμβασμό, ο προϊόν είναι συμβασμό, ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Κάθε προπολογισμό είναι προϊόν συμβασμού. Αυτοί που είχαν και τι ευθύνε από ε, κατάρτιση εθνικών προπολογισμών θα το ξέρουν καλύτερα ότι δεν ήταν εύκολο, δεν ήταν διαγωνισμό καλονή, δεν ήταν βόλτα στο πάρκο, ήταν ένα σκληρό συμβασμό. Και έτσι εδώ έχουμε ένα συμβασμό μεταξύ εθνικών συμφερόντων και γενικού καλού. Ένα συμβασμό μεταξύ εκείνων που προάγουν τη λεγόμενη πολιτική δημοσιονομικής εξυγίανσης, εξυγίανσης του προπολογισμών, κάποιοι την ονομάζουν και πολιτική λιτότητας, και εκείνων οι οποίοι προασπίζονται μια πολιτική ανάπτυξης και ε, απασχόλησης. Εγώ φρονώ ότι έχει βρεθεί ε, ο συμβασμός μεταξύ των διαφορετικών αυτών τάσεων. Και βεβαίως διαγράφεται μια στρατηγική μέσα σε αυτόν τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Μια στρατηγική γιατί, διότι θέλουμε ταυτόχρονα και να μειώσουμε βεβαίως το ε, ύψος των ε, δαπανών, όπως άλλωστε γίνεται και στα περισσότερα κράτη-μέλη. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε να προβάλλουμε εκείνες τις δαπάνες που μπορούν να φέρουν προσθέμενη αξία. Δαπάνες οι οποίες προάγουν μια πολιτική ανάπτυξης, απασχόλησης και, και καταπολέμησης της φτώχειας τόσο μέσα όσο και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει και κοσμοθεωρία, φιλοσοφία δηλαδή, αλλά και στρατηγική που στηρίζει αυτή την επιλογή, αλλά βέβαια πρέπει κανείς να διατηρήσει τις φιλοσοφικές του επιλογές, έστω και σε δύσκολες και άχαρες συνθήκες. Ας μην ξεχνάς λοιπόν αυτή η εσφαλμένη αντιπαράθεση. Δεύτερον, ο προπολογισμό αυτός δυστυχώς αντιστοιχεί στο 1% του ΑΕΠ των κρατών. Ακόμα και εκείνοι που είναι πολύ φιλόδοξοι για την Ευρώπη, δεν άκουσα ποτέ να διεκδικούν προπολογισμό σε ύψος του 1,5-2% περιοριζόμαστε μόνο σε μια συντηση μεταξύ 1,1, 1,4 το πολύ. Δηλαδή για ένα περιθώριο το οποίο δεν θα μπορούσε το άλλους να μας φέρει σε κατάσταση διχασμού. Βεβαίως και εγώ θα ήθελα όπως πολλοί από εσά ένα προπολογισμό πολύ πιο μεγάλο, πολύ πιο υψηλό. Αλλά και μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορέσετε να καταλήξετε συμφωνία για προπολογισμό σε ποσοστά διπλάσια από αυτά που έχει τώρα σχέση με το ΕΠ. Άρα λοιπόν πρέπει η συζήτηση να εντοπιστεί εκεί που ακριβώς πρέπει να πραγματοποιηθεί, στο σωστό τη πλαίσιο δηλαδή. Και με 1% του ευρωπαϊκού προπολογισμού δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα τη φτώχεια, τη ε, ανάπτυξη τη απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια συμβολή μπορεί να προσφέρει μόνο ο Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Μια συμβολή στην ε, μάχη στην οποία θα πρέπει να αποδειθούν τα διάφορα επίπεδα και κυρίω στο εθνικό επίπεδο, εκεί δηλαδή όπου υπάρχουν τα κονδύλια, έστω και σε περίοδους δημοσιονομικής εξυγίνησης. Δεν είναι αντικυκλικό μέσον ο ευρωπαϊκός προπολογισμό. Πώ θέλετε λοιπόν να φέρει αποτελέσματα αντικυκλικά, ένα ποσοστό του ε, του 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, και ακόμα και θα μπορούσαμε να συστήσουμε και τις αντικυκλικές ε, επιδόσεις άλλων ε, προπολογισμών, των εθνικών Άρα λοιπόν, μην ε, ξεχνάμε το ευρύτερο πλαίσιο. Ας μην μιλάμε σε, ε, σε δυσανάλογους όρους. Σας τα λέω απλά για να μπορώ σας επανατοποθετήσω στο γενικότερο πλαίσιο. Κάποιες ε, παρατηρήσεις που ακούστηκαν, δεν μιλάμε για νούμερα, μιλάμε για στρατηγικές. Ναι, σας το είπα. Εδώ το, τον προπολογισμό αυτόν τον χαρακτηρίζει μια στρατηγική. Το να μιλάμε για προπολογισμό όμω χωρί να αναφέρουμε αριθμητικά στοιχεία είναι σαν να μιλάμε για μια μπειραρία στην οποία δεν σερβίρεται μπύρα. Δίνουμε λοιπόν ε, νούμερα και εξηγούμε και εσείς μπορεί να απαντάτε ότι τα έχουμε ξαναδεί αυτά, περσινά ξανά στα φίλια, έχουν ξανασυμβεί. Πολύ καλά. Υποβιβάστε τα όλα αν θέλετε. Αλλά όταν μιλούμε για ανταγωνιστικότητα, όταν μιλούμε για ε, ανάπτυξη, για ε, απασχόληση και αύξηση στο σχετικό κεφάλαιο κατά 37%, 37% σε σχέση με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο που είχαμε μέχρι τώρα, μέχρι το 2013. Δεν είναι μηδενικό, δεν είναι copy-paste, δεν είναι απλή αντιγραφή και περσινάξινα στα φίλια. Είναι μια τεράστια αύξηση της πρικοδότησης και εδώ πέρα πιστεύω θα πρέπει κανείς να διατηρήσει και μια στις αναλογίες, να ξέρουμε γιατί μιλάμε και τι συγκρίνουμε. Είναι αντικοινωνικός ο προϋπολογισμός, στρέφεται κατά της κοινωνίας. Μα έχει αυξηθεί το μερίδιο για τα πιο φτωχά κράτη από το Ταμείο της Συνοχής. Έχει αυξηθεί το σχετικό, η, η αναλογία δηλαδή, ε, για εκείνους που έχουν πιο πολύ ανάγκη και έχει παραμείνει και έχει ενισχυθεί επιπλέον το, το πρόγραμμα για του πιο φτωχού, όπω περιγράψε και ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε διατηρήσει το πρόγραμμα στην, για τη βοήθεια στην ανάπτυξη. Έχουμε διατηρήσει του στόχου τη χιλιετηρίδα. Έχουμε εισαγάγει ένα νέο πρόγραμμα που βρίσκεται στην τελική φάση των διαπραγματεύσεων τώρα για 6 δισεκατομμύρια ευρώ ε, που θα στηρίξουν τους νέους ανέργους. Πρόκειται για ένα προπολογισμό με οικονομική στρατηγική και εδώ παραπέμπω στο 30% που σας ανέφερα τώρα, είναι ένας προπολογισμό που έχει κοινωνικό χαρακτήρα, μεταξύ άλλων. Τώρα και στα άλλα θέματα, διαφορά, αποκλήσει μεταξύ των πιστώσεων υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών. Ε, θα σας ε, παραπέμψω και στην εμπειρία που έχω ως ε, υπουργό Αρμόδιος για τα δημοσιονομικά στη χώρα μου. Πάντα είχαμε αποκλήσεις μεταξύ πιστώσεων πληρωμών και πιστώσεων υποχρεώσεων. Ιδάλλον δεν θα, χρειάζεται, δεν θα χρειαζόταν να υπάρχουν ε, πιστώσεις υποχρεώσεων. Γι' αυτό υπάρχουν. Και θα σας αναφέρω τα Το 2005 και δεν θα μιλήσω όπως ο συνάδελφος και φίλος. Το φίλος ε, για λόγους αυρότητας και μόνο το αναφέρω. Χωρίς όμως να θέλω να προσωποποιήσω τη συζήτηση, γιατί εγώ δεν ήμουν εδώ το 2005, δεν ήμουν εδώ. Άλλο ήταν ο Πρωθυπουργό, ξέρετε, έχετε ακουστά. Οι διαφορές λοιπόν μεταξύ των πιστώσεων υποχρεώσεων και των πληρωμών στη χώρα μας ήταν της τάξης του 5,4% και από ό,τι έμαθα, μάλιστα ποτέ δεν έχει γίνει και σχετικό διάλογο για το θέμα αυτό. Και τώρα είμαστε στο 5,7%. Αλλά τι με τόσο συνέβαιναν πριν από 7 χρόνια. Ο, ο διάλογο έγινε κατά πολύ συγκεκριμένου όρου και με την επιμελητιακή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το πώς μπορούμε να καλύψουμε το χάσμα μεταξύ πιστώσεων πληρωμών και πιστώσεων υποχρεώσεων. Υποχρεώσεων πρώτα πληρωμών μετά. Ε, και επίσης, αν κάνουμε το έθρισμα των πιστώσεων υποχρεώσεων στην επταετία που έχει μόλις ε, εκπνεύσει, φτάνουμε στα 991. Ε, ξέρετε, 91 ή 91 λέμε στα γαλλικά, ε, ανάλογα με τον είναι κανείς Βέλγος ή Γάλλος, σε περιπτώσει 991 το ίδιο είναι το νούμερο, δεν αλλάζει τίποτα. Εάν, μάλιστα, εάν δε αφρίσουμε τις πιστώσεις πληρωμών που ενέκρινε το Συμβούλιο μαζί με το Κοινοβούλιο, ξεπερνούμε το 100 δις λιγότερα, δηλαδή 875. 875 σε πιστώσεις πληρωμών αντί για τα 991 στις υποχρεώσεις. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά λοιπόν, ε, γιατί διαφορές και αποκλήσεις υπήρχαν πάντα. Η κύρια διαφορά όμως τώρα είναι ότι έχουμε ε, μηχανισμό ευελιξία, ο οποίο καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, κάνει το maximum possible όπω λέμε τόσο ωραία στα αγγλικά και βεβαίω θα πρέπει να συστήσουμε ει βάθος για το πώ θα λειτουργήσει και θα συνεχιστεί ο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα τρίτο στοιχείο. Πιστώσει πληρωμών τη περίοδου του προηγούμενου δημοσιονομικού πλαισίου. Τα 875 δισεκατομμύρια είναι ακόμα λιγότερα από αυτά που έχουμε προτείνει τώρα, τα 908 δηλαδή, που, είχαμε, που έχουμε προτείνει τώρα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το προσχέσιο δημοσιονομικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα 33 λιγότερα. Άρα μπορούμε να το διαχειριστούμε το ζήτημα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τελευταίο στοιχείο. Βεβαίω θα πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση. Το είπα επανελειμμένο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και αυτέ τι 30 ώρε που κράτησαν οι συζητήσει μα, το συζητήσαμε, το είχαμε άλλωστε συζητήσει και τον Νοέμβριο. Είπαμε πρέπει να εξασφαλιστεί συμφωνία για τα 27 κράτη-μέλη. εκ εκτρώνουν κάνευ. Και εκτρώνουν κάνευ σημαίνει ότι πρέπει να συνεχίσουμε μετά. Δεν κλείνει εκεί η διαδικασία. Πρέπει να συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση και άρα να βρούμε λύσει, ανοίγματα μεγάλα ανοίγματα, σημαντικά ανοίγματα στον, στην ευελιξία, στους ιδίους σπόρους στην ενδεχόμενη αναθεώρηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι την ειδικόνη ως ε, στις προτάσεις για την ε, αναθεώρηση. Βέβαια, θα πρέπει να συζητήσουμε τις διατυπώσεις, γιατί πάντα πολλές είναι διατυπώσεις να μην ε, αναθεώρηση. Αλλά παρακαλώ όλους τους Ευρωπαίους να καλοσκεφτούν και να σκεφτούν πολύ προσεκτικά τι συνέπειε μπορεί να έχει μια διαδικασία ενιαύσεων προπολογισμών. Γιατί? Γιατί τότε δεν θα αφήσετε καμία προοπτική για όλους αυτούς που έχουν στρατευθεί στην έρευνα και την ανάπτυξη, για όλες αυτές τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που μας ζητούν, απαιτούν προοπτικές, για όλους αυτούς τους άνεργους νέους, για όλους αυτούς που έχουν αποθέσει τις ελπίδες τους αυτούς τους κρίσιμους τομείς. και τα κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Σας παρακαλώ λοιπόν να το καλοσκεφτείτε και να δράσετε υπεύθυνα για να μην περιπέσουμε στους ε, νεάφρους Το copy-paste τότε θα συμβεί, για όσους επισήμαναν ε, στην παρατήρηση. Για τότε μεταρρύθμιση θα γίνεται. Θα έχουμε περιμείνει στα κονδύλια στις πιστώσεις του 2013 και απλώς θα συνεχίζουμε τη λειτουργία των γραμμών εκείνων του προπολογισμού που χαράχθηκαν πολλά χρόνια πριν. Η πολιετής προπολογισμοί, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δίνει προοπτικές για το μέλλον ο ενιάξιος προπολογισμό μας φέρνει σε συζητήσεις με δεδομένα μόνο ετήσια, οδηγεί σε ε, απώλεια πολλών πόρων, ενέργειας, προσπαθειών, κόπων για ένα αποτέλεσμα πολύ ισχνό, ένα πολύ περιορισμένο προπολογισμό. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, λοιπόν, αυτός ο πολιετής προπολογισμό, είναι ένα σημαντικό πολιτικό ε, εργαλείο, ε, ενσωματώνει μία πολιτική επιλογή, μια στρατηγική επιλογή. Ξέρω ότι πολλά στοιχεία του σας φέρονται άχαρα και δεν έχω ε, καμιά επιφύλαξη να δεχθώ τις επιλογές σας και την κριτική σας αυτή. Από την όλη όμως, για να μην περιπέσουμε σε μια πολύ πιο σοβαρή κρίση, παρακαλώ να είστε πολύ προσεκτικοί και να δράσετε με τρόπο υπεύθυνο. Ευχαριστώ. Θα ζητήσω από τους συναδέλφους που θέλουν να λάβουν τον λόγο να τηρήσουν ρητά το χρόνο που έχουν, διότι ε, πρέπει να φύγει και ο πρόεδρος που εδώ πάει. Ο κύριος Στάσεν, για, η κυρία Στάσεν, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, θα είμαι σύντομη και περιεκτική. Ακούσαμε όλη αυτή τη τεχνική επεξήγηση. Η αλήθεια όμως ποια είναι. Ελαστικότητα για 7 χρόνια. Πώς θα εφαρμοστεί αυτή. Και ο Σούλς το είπε Μίλησε για τα 16 εκατομμύρια προς τις χώρες με τη διαφορά που υπάρχει. Είναι σαν να έχει πτωχεύσει βασικά η Ευρώπη. Και θέλω να πω ότι είναι σκανδαλώδες που ζητάμε εδώ μυστική ψηφοφορία. Είναι ύβρις προς την δημοκρατία αυτό. Ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Η κυρία Λιωτάρ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φανουρομπάου. Εδώ ακούσατε ε, τις διαμαρτυρίες μας και εσείς ε, βέβαια μείνεστε του σχεδίου σας. Αλλά είπαμε ότι δεν πρόκειται μόνο για τα νούμερα, πρόκειται για την αδυναμία του σχεδίου αυτού να στηρίξει τους πιο αδύναμους, ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης. Εμείς θέλουμε τα χρήματα να πηγαίνουν κατευθείαν στον Ευρωπαίο πολίτη και όχι μέσω άλλων προγραμμάτων από τα οποία τελικά δεν θα μπορέσουν οι πολίτες και οι πιο αδύναμοι να αποφεληθούν. Ο κύριος 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Επιτροπή και το Συμβούλιο για την απόφαση που λάβανε. Γιατί θα πρέπει να επισημάνω ότι μπορεί να χαίρομαι για την ε, ε περικοπή των κονδυλίων στο με τα οποία θα συμβάλλει η Δανία και γενικότερα την τάση για πιο προσεκτικό η συγκατάρτιση του προπολογισμού. Αλλά νομίζω ότι εν γέννη δεν έχει βρεθεί λύση για το πιο σοβαρό πρόβλημα που είναι το ατέρμον αυτό πήγαινε λέει, μεταξύ Βρυξελών και Στρασβούργου. Δεν έχουν δοθεί λύσεις για τα ερχοτικά ταμεία και τους σπόρους που αυτά απορροφούν. Βλέποντας ε, το περιεχόμενο αυτής της ε, συμφωνίας, πρέπει να πω ότι έχουμε από τη μια 27 δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις, Μπορεί να μην με βρίσκουν όλε συμφωνώ, αλλά παντό είναι δημοκρατικά εκλεγμένε, οι οποίε είναι υπόλογε ενώπιον των εθνικών του κοινοβουλίων και οι οποίε μπόρεσαν να καταλήξουν μέσα στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε ένα συμβασμό. Και από την άλλη έχουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο δεν εκπροσωπεί το μισό ευρωπαϊκό προπολογισμό και δεν έχει καν το θάρρο να αρθεί στο περιστάσεων και να εξηγήσει σε τι μπορεί να εξυπηρετεί ένα ευρωπαϊκό προπολογισμό και, τι, και πού πηγαίνουν τα κονδύλια. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ευθύνε του κυρίου Μπαρόσο, που δεν εκπροσωπεί ούτε το μισό πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα από τις ε, δημοκρατικά εκλεγμένες κυβερνήσεις. Ο κύριος Κάλλαν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Δεν ξέρω αν υπάρχουμε στην κατηγορία των καλών ή κακών Ευρωπαίων σύμφωνα με τον κύριο Παναδομπάη. Να πω κάτι που κανείς άλλος δεν έθεσε. Την ε, θετική άποψη για την ε, Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Η Συμφωνία για την... Ε, η συμφωνία αυτή θα, έκανε πολύ καλύτερα, ε, θα πολύ καλύτερα αποτελέσματα για τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη από ότι όλες οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Όλοι θέλουμε βελτίωση στον προπολογισμό και χάρηκα που και εγώ θα ήθελα να υπάρχουν μικρότερες δαπάνες στη γεωργία, στη διοίκηση. Στην πραγματικότητα θα γίνουν διαπραγματεύσεις. Φαντάζομαι ότι το Κοινοβούλιο εν τέλει θα υπερψηφίσει τη συμφωνία γιατί η εναλλακτική λύση οποιοδήποτε άλλο προπολογισμό θα ήταν χειρότερη αν μη τι άλλο, αλλά αυτό που θα ήταν γελίο είναι να καταψηφίσουμε ε, με μυστική ψηφοφορία. Αυτό θα ήταν πραγματικά γελίο, πρέπει, πρέπει να γίνει δημοσία. Δεν θα ε, χρειαζόταν να γελιοποιήσουμε το Κοινοβούλιο ανά την Ευρώπη με μυστική ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντουιρόν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Τέσσερι παρατηρήσει, Πρώτον, ναι, μπορεί να ζήσουμε χωρίς πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχουν οι τεχνικές και νομικές ρυθμίσεις σχετικά. Δεύτερον, η φιλοσοφία του πλεχτού σα δεν είναι ξεκάθαρη. Εγώ δεν την κατάλαβα, ούτε και θέλω να καταλάβω ποια είναι η φιλοσοφία σας. Τρίτον, η πολιετή ε, δέσμευση ανατμήμα σε πολιετή πολιτές πλαίσιο δεν στέκει. Δεν μπορεί να μας πείτε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν πολιτή προγράμματα γιατί δεν έχουμε πολιτές ε, προϋπολογισμό. Λοιπόν, τώρα, μειώνετε τις ε, πληρωμές την ώρα που μειώνεται και τις υποχρεώσεις. Μιλάτε για 37%, ξεχνάτε όμως να πείτε ότι ξεκινά από ένα δημοσιονομικό προπολογισμό που κόβουμε 24% σε σχέση με, τον με την πρόταση προπολογισμού της Επιτροπής, όπου ήταν ήδη περικομμένος. Πραγματικά, ξανασκεφτείτε το, ξανά ξανασκεφτείτε το, πριν υιοθετήσετε την τελική σας θέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερχόφστατ, ένα λεπτό. Ναι, δύο σημεία. Πρώτον, τα ποσά με τους αιτήσους προπολογισμούς θα είναι τα ίδια. 15 δις για το 2013, 15, 15,6 για το χρόνο. Θα είναι ακριβώ το ίδιο ποσό εάν πάμε σε νέα στου Εδώ τα έχω. Το δικό σα παράρτημα είναι στα συμπεράσματά σα, δεν το βλέπετε. Ακριβώ τα ίδια με τον προπολογισμό του 2013. Άρα δεν έχει καμία σημασία για τον, το αν θα έχουμε νιάυσιο ή μη. Δεύτερον, ε, υπάρχει ένα διαρκές πρόβλημα διονγκούμενου ελλείμματος, χρέους. Μπορεί να μου λέτε ναι, θα και τα λοιπά. Όχι διονγκούται διαρκώ, και γι' αυτό άλλωστε και ζήτησα, ο κύριε Πρόεδρε, την ΑΔΕ, γιατί δεν επιτρέπεται κανονικά, να διανύμω το σχετικό έγγραφο στο οποίο καταγράφω πω διονγκούται το χρέο. 60 δι το 2000, τώρα είμαστε 200 δι και θα προχωρήσουμε στα 300 πριν καταλάβουμε καλά καλά τι έχει γίνει αυτό το μεγάλο έλλειμμα, το οποίο προκαλεί πάλι και το ενισχύει ακόμη αυτό το ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Παρακαλώ λοιπόν τους κλητήρες να διανύμουν στη συνέχεια για να δούνε τι συνέπειες έχει για το έλλειμμα το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Κάλφιν, τέσσερα λεπτά. δεν αμφισβητώ τις Φιλοευρωπαϊκέ σα απόψει. Αλλά αμφισβητώ ότι το κατά πόσο ο προπολογισμό που εγκρίθηκε είναι φιλοευρωπαϊκό. Το θέμα δεν είναι να παίζουμε με τα νούμερα. Αυτό που πετύχατε είναι ότι βρήκατε τον ελάχιστο κοινό παρονομαστή που περιέργω είναι αρεστό σε κάποιους κύκλους που θέλουν να στραγγαλίσουν τις ευρωπαϊκές πολιτικές πριν η χώρα τους εγκαταλείψει την Ένωση. Αυτό ήταν η βάση του συμβιβασμού που είδαμε. Οι αντιδράσει από τι πολιτικές ομάδες στο Κοινοβούλιο είναι εύγλωτε. αν δείτε ποιο μιλάει και τι λέει. Είπατε ότι είστε ανοιχτοί για συζητήσεις βάσει στοιχείων. Ναι. Αλλά ε, η άνοιξη, η, αύξηση μπορεί να προκύψει, θα προκύψει μόνο αν περάσουμε ε, κονδύλια από τη συνοχή στην κατηγορία 1. Μπορώ να σας δώσω τα στοιχεία του ΩΣΑ για τις δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη. Δεν το κάνω, ωστόσο γιατί θα το, μπορείτε να το κάνετε. Θα δείτε ότι οι χώρες το 2010 δαπανούν μεταξύ 60 και 100 περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιαπωνία, ολόκληρη την Ένωση, η Ιαπωνία, Κορία, Κορέα, Ισραήλ, Ηνωμένε Πολιτείε. Θα έχουν περισσότερες δαπάνες. Το 2020 θα μιλήσουν ακόμα περισσότερο. Δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι, θα αυξάνει, ότι αυξάνει ο υπολογισμό. Αυτό δεν στέκει. Μιλάτε για την ανεργία των νέων. Όντω, ε, εξαιρετική λύση. Δείτε όμω τα νούμερα. Τρία δι. Τα άλλα τρία προέρχονται νέα. Τα άλλα προέρχονται από το υφιστάμενο κοινωνικό ταμείο. Θα σα δώσω κάποια άλλα στοιχεία για τα νέα κράτη-μέλη για να διατηρήσουν την ε, ε κατάσταση βάσει του σουηδικού μοντέλου χρειάζεται 21 δις το χρόνο. Στην Ευρωζώνη μόνο. 13 δις συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο προπολογισμό της Ένωσης θα δαπανίσει 6 δις σε 7 χρόνια. Τι αντίκτυπο θα έχει αυτό. Ωραία να μιλάμε για την, ενεργία, για την καταπολέμηση της ενεργείας των νέων, για πολιτικές, αλλά όταν βλέπουμε τον αντίκτυπο αυτών των κονδυλίων θα δείτε ότι δεν λειτουργεί. Το ίδιο και με τη συνοχή. Υπάρχει σαφής μείωση των πόρων ε, συνοχή, καθαρή μείωση των πόρων για τη συνοχή με περισσότερους δικαιούχου. Η ευρωπαϊκή οικονομία και οι περιφέρειες θα έχουν μεγαλύτερη συνοχή. Πώς το λέτε αυτό, δεν μπορείτε να το πείτε. Τέλο, πρόεδρε. Είναι σαφές και το είπατε. Δεν είναι δυνατό δεν είναι αναγκαίο μάλλον να έχουμε περισσότερη Ευρώπη έχοντας υποχρεωτικά και περισσότερα χρήματα. Ότι περισσότερη Ευρώπη δεν σημαίνει περισσότερα χρήματα. Λιγότερα, χρή, ε, λιγότερα χρήματα ωστόσο σημαίνει λιγότερη Ευρώπη. Και αυτό βλέπαμε με τον προπολογισμό. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Κάποιοι θα το θέλαν. Βεβαίω. Θέλουν να δουν λιγότερη Ευρώπη. Δεν είναι όμω αυτή η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Διότι όντω θα θέλαμε να υπάρχουν ευρωπαϊκέ πολιτικέ. Μιλάμε για ευελιξία. Μπορούμε να έχουμε ευελιξία αν έχουμε πόρου. Εσεί και ο πρόεδρο Μπαρόζο μιλάτε για την ευελιξία μέσα στα αίτια, αλλά αν έχετε πολύ χαμηλέ πληρωμέ, δεν θα έχετε τίποτα να μεταφέρετε από χρόνο σε χρόνο. Απλά θα ξαναπηγαίνετε στη θέση της ομοφωνίας όπου κάθε χώρα μπορεί να μπλοκάρει οποιαδήποτε απόφαση στον προπολογισμό. Και αυτό γίνεται. Εμεί δεν το λέμε αυτό ευελιξία. Μιλάτε για διαδικασίες ομοφωνίας που πρέπει να είναι ευέλικτες. Ναι, το παρατρύνουμε αυτό. Αν θέλουμε να έχουμε ευελιξία πρέπει να έχουμε λιγότερη ομοφωνία στο Συμβούλιο. Και αυτό πάει μαζί με την ευελιξία. Και προς τα εκεί πρέπει να στραφούμε. Αλλιώς λέμε ωραία λόγια, μιλάμε για ευρωπαϊκές δεσμεύσεις, αλλά δεν έχουμε τα μέσα για να υλοποιούμε αυτά που υποσχόμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τελευταίο αγορητής, ο κύριο Μπέγκε, πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώντας, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με τον κύριο Κάλφιν και θα ήθελα να πω ότι ο ενθουσιασμός με τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι μάλλον περιορισμένος. Ένα πράγμα όμως καταλάβανε, από ό,τι φαίνεται, για τη θέση του Κοινοβουλίου ότι εάν δεν ήμουν ικανοποιημένο το Κοινοβούλιο από τα αποτελέσματα, υπάρχουν και εναλλακτικέ. Η προειδοποίηση ότι μπορεί να οδηγηθούμε σε ένα σενάριο πολύ χειρότερο και πολύ κακό εάν δεν συμφωνήσουμε είναι ατυχής και αβάσιμη. Όχι. Έχετε βολευτεί σε αυτήν την κατάσταση. Το, το Συμβούλιο επιλέγει και ότι το Κοινοβούλιο αναγκάζεται να παρακολουθήσει. Όχι, μπορεί το Κοινοβούλιο να αντιδράσει και να καταλήξουμε σε ενιαύτους προπολογισμού. Και επίση θα ήθελα να πω πώς καταλήξατε κύριε Πρόεδρε, εδώ πέρα ανέφερε ο συνάδελφο τα αποτελέσματα για την έρευνα. Χρειάζεται να δώσουμε στην Ευρώπη μια μεγάλη όθηση και είτε πρόκειται για ευρωπαϊκό προπολογισμό και προσπάθειες ε, των επιχειρήσεων, είτε πρόκειται για εθνικούς προϋπολογισμούς η Ευρώπη χρειάζεται συνολικά πάνω από 120 δισεκατομμύρια το χρόνο. Καλό λοιπόν να τα λέτε στα σχέδια, αλλά δεν αρκούν για να αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές προκλήσεις. Και θα ήθελα να επισημάνω το εξή επιπλέον. Ο κ. Λαμασούχ, πρόεδρο τη Επιτροπή των Προπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και προ τον επικεφαλή ε, του επιτελείου σα, κ κ. Φαν Ρόμποϊ απέστειλε μια επιστολή λέγοντας ότι 64, σελίδε σελίδες των συμπερασμάτων ε, δεν έχουν ε, δεν, γράφουν, δεν καταγράφουν το πνεύμα αυτό το ευρωπαϊκό το οποίο θα κερδίσει τον πολίτη της Ευρώπης και δεν έχουν σημασία τα 5-10 εκατομμύρια πάνω κάτω. Έγραφα λοιπόν και προτάσεις όπου καταγράφεται για τα κράτη-μέλη και το εθνικό τους ακροατήριο του, το, τι είδου ε, συνέπειες μπορεί να έχει μία ή άλλη επιλογή τα τόσα ή τα τόσα εκατομμύρια στην γεωργία ή στη συνοχή σε κάποιο άλλο αλλά δεν κοινοποιούνται σε εμάς ε, με υποχρεώνω να σας πω απερίφραστα ότι είτε θα μας κοινοποιήσετε τα ίδια στοιχεία, είτε δεν θα συνεργαστούμε πλέον. Απαιτούμε την ίδια διαφάνεια, απαιτούμε την ίδια ενημέρωση, ώστε να μπορώ και εγώ να λαμβάνω τις αποφάσεις μου γιατί το σκάνδαλο δεν είναι το να ζητούμε μυστική ψηφοφορία, αλλά το να υπάρχουν ε, συζητήσεις και ξεμένων των θυρών στο Συμβούλιο, χωρίς καμία διαφάνεια, χωρίς να γνωρίζει ο πολίτης περί τίνος πρόκειται και τι διακυβεύεται. Αυτό είναι το πραγματικό σκάνδαλο. Εάν δούμε λοιπόν ε, τα όσα είναι τη σοφία του έχει αποφασίσει για την έρευνα και την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Συμβούλου, για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, για την ιστορική και εξωτερική ασφάλεια, για το ρόλο της Ευρώπης ανά τον κόσμο, Όλα αυτά δεν συνάδουν με τα νούμερα που μας παρουσιάσατε. Κάπως θα πρέπει να τα παρουσιάσετε στις ε, διαπραγματεύσεις και γι' αυτό καλό θα είναι να ε, εγκαταλείψετε τις πολιτικές αυτές προτεραιότητες οι οποίες δεν ευθυγραμμίζονται με το πολιτές νοσονομικό πλαίσιο. Τα ραλ, τα υπόλοιπα προς ε, εκαθάριση. Και αυτά συζητήθηκαν βεβαίως. Εάν δεν καλυφθούν τα ποσά, θα παραμένουν κονδύλια μέχρι την περίοδο μετά το 2020, πράγμα το οποίο θέλουμε να αποφύγουμε. Πρέπει να βρούμε έναν τροπικό, διαφορετικό τρόπο να ε, ρυθμίσουμε το ζήτημα των υπόλοιπων προς εκαθάριση και να εκαθαρίσουμε έτσι τον προϋπολογισμό ώστε να μην αντιμετωπίσουμε τα ίδια προβλήματα, το, την ίδια φύρα ουσιαστικά ε, ή το ίδιο έρμα καλύτερα στον επόμενο, στο επόμενο πολιτής δημοσιονομικό πλαίσιο. Ευελιξία, ήδη οι πόροι, ε, εδώ χρειαζόμαστε λύσεις ευέλικτες, ενδεχομένως και με προτάσεις για περισσότερους ιδίους πόρους. Ευελιξία σημαίνει ευελιξία για τους πάντες, για κάθε είδους υποχρέωση, για κάθε είδους πληρωμή. Αυτό σημαίνει ευελιξία. Προς κάθε κατεύθυνση. Και στη συνθήκη τη Λισαβόνα, σα υπενθυμίσω ότι είχε γίνει λόγο για ευελιξία, χωρί την οποία δεν θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε, να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε το Γαλιλαίο. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι στα συμπεράσματα να ανοίγει η θύρα για την ευελιξία, αλλά προφανώ δεν επαρκεί αυτό το μικρό άνοιγμα. Και κύριε Φεγόφστα, θα ήθελα ξεκάθαρα να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει το νέο κοινοβούλιο αυτό να έχει την ε, ε, δυνατότητα να εγκρίνει την ε, νέα αυτή συμφωνία. Οτιδήποτε άλλο θα αποκλίνει πολύ από τη δημοκρατική νομότητα. Για δε τους δύο σπόρους. εδώ υπάρχει μια ρήτρα ότι θα πρέπει να την εξυπήσουμε και πρέπει τα κράτη-μέλη να, μετακινηθούν ως προς τις θέσεις τους και να, να δώσουν νέες λύσεις για χρηματοδότηση. Για δε τη δυνατότητα διατύπωσης δικών μας προτάσεων, το δημοσιονομικό πλαίσιο, πώς θα το βλέπατε. Ε, εμείς είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε, είμαστε έτοιμοι, έχουμε προετοιμαστεί, έχουμε κάνει τη δική μας δουλειά και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι είμαστε διατεθειμένοι ακόμη και να φτάσουμε στην έγκριση μιας τελικής συμφωνίας μόνο όταν θα είμαστε βέβαιοι για την ποιότητα και το περιεχόμενο των πολιετών ε, προγραμμάτων. Μόνο όταν γνωρίζουμε ότι υλοποιούνται οι στόχοι μας, ότι εξασφαλίζονται οι προτεραιότητες μας και ότι και η πολιτική η γεωργική αλλά και η πολιτική της έρευνας θα χρηματοδοτηθούν επαρκώς, θα καταλήξουμε συμφωνία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Μπαρός. ευχαριστώ όλους τους παρόντες. Πέρα στην εδριά σας.